Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ε, χαιρετίζω σήμερα το πρωί. Βλέπετε ότι δεν είναι εδώ ο Μάλκολ Χάρμπορντ. Με παρεκάλεσε ε, να τον αντικαταστήσω γιατί είναι σε κάποιο συνέδριο και ε, επίσης απουσιάζουν όλοι οι αντιπρόεδροι. Πιστεύω ότι παρόλα αυτά θα κάνουμε καλή εργασία και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Πράγμα το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε μια καλή συζήτηση διότι ότι αν δεν έχουμε πολλούς συμμετέχοντες θα έχει περισσότερο χρόνο κάθε συμμετέχον. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι εχθές στην ε, ε, συνεδρίαση των συντονιστών συζητήσαμε ε, για την πρώτη την πρώτη ε, εξέταση ε, των προτύπων και αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη συζήτηση σε μία ανάγνωση γιατί το Συμβούλιο είναι έτοιμο να μας προσεγγίσει και στη συνέχεια ε, για τους δύο φακέλους που έχουμε προσυζήτηση θα τους ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Ε, όπως ξέρετε χρειαζόμαστε μια ε, ψηφοφορία με 21 ε, θετικές ψήφους για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία. Αυτό προς ενημέρωσή σας. Σας υπενθυμίζω και πάλι πριν θα σας το μάλλον ξανά υπενθυμίσω πριν ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες κατά τρόπον ώστε να το γνωρίζουν και όσοι συνάδελφοι δεν παρίστανται αυτή τη στιγμή. Ξεκινάει λοιπόν η, πρώτη, η συζήτηση του πρώτου θέματος και με στενοχωρεί διότι σήμερα δεν είμαι ε, μόνο πρόεδρος αλλά εκτελώ και χρέη συντονιστή και χρέη συγκητή. Οπότε ε, θέλω να ε, αναφερθώ στην έκθεση ε, για την πρόσβαση στις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες. Δεν, δεν θα συνυπολογίσω ποιος δεν είναι εδώ από τους σκιώδεις εισηγητές γιατί ενδεχομένες μπορεί να έρθουν εντωμεταξύ αλλά πρέπει να προχωρήσουμε και σας υπενθυμίζω ότι έχουμε ε, το web streaming, τη μετάδοση στο διαδίκτυο και γι' αυτό το λόγο όλοι οι ακροατές μας και οι θεατές μας που ενδιαφέρονται για την εργασία μας θα πρέπει να μπορούν να παρακολουθήσουν στον προβλεπόμενο χρόνο. Για την ε, έκθεση την οποία ε, έχω υποβάλει εδώ έχουν υποβληθεί 27 τροπολογίες τις οποίες θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και οι περισσότερες ακολουθούν μία κατεύθυνση ε, σύμφωνα με την οποία δεν είναι δύσκολο να τη συζητήσουμε και γενικώ λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποβλέπει τα κράτη-μέλη ε, ε, υποχρεωθούν να έχουν πρόσβαση ε, σε έναν ουσιαστικό τραπεζικό λογαριασμό όπου μπορεί να κάνει κινήσεις ε, για τα χρήματά του. Υπάρχει διαφορά σε διάφορες χώρες. Ε, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία το ίμιση των κατοίκων δεν έχουν δυνατότητα προσβάσεως τραπεζικό λογαριασμό. Το ίδιο ισχύει και στη Γερμανία για περίπου 3 εκατομμύρια πολιτών και ως εκ τούτου εδώ θα ήθελα να τονίσω και πάλι ε, κατόπιν των συζητήσεων που έχουμε κάνει ότι είναι ε, το δικαίωμα σε έναν τραπεζικό λογαριασμό δεν είναι θέμα υποχρεώσεως εάν δεν τον θέλει ας μην τον ε, αποκτήσει αν είναι άστεγος, αν δεν έχει επαρκή χρήματα, ε, αν είναι ένας φοιτητής σε μία άλλη χώρα, τότε ε, μπορεί να κινηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που θέλουμε είναι να διευκολύνουμε αυτές τις κινήσεις. Εχθές συζητήσαμε το θέμα με τους συναδέλφους συντονιστές για να μπορέσουμε ε, να συζητήσουμε τις 87 τροπολογίες και εντωμεταξύ Έχουμε 10 ε, συμβιβαστικές ε, επί τις οποίες επιφυλασσόμαστε ε, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων και θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στα πιο βασικά θέματα. Το πρώτο θέμα είναι το κόστος, δηλαδή τι μπορεί κανείς να απαιτήσει από τους πολίτες όπου έχουν έχω λάβει πάρα πολλέ τροπολογίες ε, οι μεν λένε ότι δεν πρέπει να υπάρχει κόστος και ποτέ θα πρέπει για πάντοτε να είναι δωρεάν και υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι ζητούν ένα ελάχιστο ποσό ε, για τις χρεώσεις και το έχουμε συζητήσει. Η δικιά μου πρόταση λοιπόν είναι να πούμε ότι κατά κανόνα οι λογαριασμοί αυτοί θα πρέπει να έχουν το ελάχιστο δυνατό κόστος, ιδίως αν υπάρχει κόστος, ε, δεν θα πρέπει να είναι τεράστιο αυτό. Ε, ε, ξέρω ότι αν μιλάμε για ένα τεράστιο με καταλαβαίνετε ε, αν εργάζεται βέβαια κανείς ε, στο γραπτό λόγο μεταξύ γαλλικών και αγγλικών και μιλά γερμανικά είναι δύσκολο να εκφραστεί με ακρίβεια ε, ε, πέραν αυτού πρέπει να δούμε πώς θα διεκπαιρεώσουμε τα θέματα αυτά κατά τρόπον ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε ένα λογαριασμό ε, η οποία θα απαγορεύεται πολύ σωστά σε περίπτωση τρομοκρατίας ή παρεμφερών αιτιών και το ερώτημα ήταν αν έπρεπε αυτό να συζητηθεί σε αυτή την έκθεση ή να παραπέμψουμε στην ισχύουσα νομοθεσία και στο τέλος συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να αναφερθούμε στην ισχύουσα νομοθεσία διότι θα πρέπει να ξέρουμε ε, τι, ε, ε, τι μπορεί κανείς να κάνει σαν επέμβαση σε ένα τέτοιο λογαριασμό για να μην μπορεί κανείς από την πίσω πόρτα να ε, ε, προκαλέσει ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή να χρηματοδοτήσει παράνομες ενέργειες. Πέραν αυτού είπαμε ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ένας βασικός λογαριασμός όταν ανοίγεται ε, δεν υποχρεώνει δεν μπορεί να υποχρεώσει τον ε, πολίτη ε, ή την ε, τράπεζα να συνδέσει με το άνοιγμα του λογαριασμού ορισμένες ασφάλειες ή ορισμένες δεσμεύσεις. Ένα θέμα όμως στο οποίο δεν έχουμε συμφωνήσει μεταξύ κομμάτων για το πώς θα το αντιμετωπίσουμε είναι το θέμα της σχέσεως που πρέπει να έχει ένα άτομο με το κράτος αν έχει ανοίξει έναν βασικό λογαριασμό. Η δικιά μου πρόταση είναι ότι σε περίπτωση τέτοιου λογαριασμού να υπάρχει μία διασύνδεση του ατόμου που έχει το λογαριασμό με ε, το κράτος και το ερώτημα είναι αν αυτό μπορεί να, είναι, μπορεί να αποδεικνύεται διότι ε, υπάρχει ο κίνδυνος να ζητείτε εκ των υστέρων μία απόδειξη και όταν ε, ε, και όταν δεν έχει κανείς λογαριασμό και δεν μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι και πας στην τράπεζα και δεν σου ανοίγει το λογαριασμό διότι δεν έχεις μία νόμιμη διεύθυνση είναι θέματα τα οποία έχουμε προσπαθήσει να λύσουμε με μία διατύπωση και με ενδιαφέρει να ακούσω τι έχουν να πούνε επί του θέματος οι σκιώδεις εισηγητές. Ένα άλλο θέμα είναι οι ε, εναλλακτικέ Δυνατότητα δυνατότητος ε, επιλύσεως των διαφορών και το collective redress ε, και ε, υπάρχει μία δυνατή διατύπωση την οποία θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει αποδεκτή και σέβεται τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που είναι επίσης βασικό να παραμείνει. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι, αλλά στην περίπτωση αυτή μπορεί να μου το υπενθυμίσουν οι σκιώδεις εισηγητές και αν έχω ξεχάσει κάτι βασικό θα επανέλθω. Τώρα όμως θέλω να δώσω τον λόγο εις τους συναδέλφους και καταρχήν στους ε, σκιώδεις εισηγητές ο Χάνς Βίντερ Μάιερ του ΕΛΚ ε, δεν παρίσταται αλλά αντικαθίσταται. Ε, από τον κύριο Έλερ. Ε, ευχαριστώ. Σήμερα το πρωί μου ζήτησε ο συνάδελφος να τον εκπροσωπήσω και μπορώ να σας απευθύνω το λόγο και γερμανικά. Μας είπατε τι θα ήταν λογικό. Μιλούσαμε για τιμές και ο κύριος Μαγιέρ μου ζήτησε να σας πω τα εξής. Ευχαριστούμε για τις συμβιβαστικές λύσεις, εκ των οποίων οι περισσότερε είναι λογικές, να υπάρχει ένας βασικός λογαριασμός δωρεάν ή με αντίστοιχο κόσος. Πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστές. Δεν πρέπει οι τράπεζες να κερδίζουν από αυτούς τους λογαριασμούς, αλλά δεν, είμαστε δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τις τράπεζες να διαθέτουν και να ανοίγουν λογαριασμούς δωρεάν. Ιδίως όταν υπάρχουν και δυνατότητες ε, πληρωμών ε, μέσω του διαδικτύου, δηλαδή ε, μέσω του web banking ή μέσω του κινητού τηλεφώνου, το οποίο όμως εμείς δεν επικροτούμε. Ο συμβιβασμός τον οποίο προτείνει ο συνάδελφος είναι ότι ότι το κόστος θα πρέπει ε, να είναι όντως αντίστοιχο του λογαριασμού και ε, ε, πρέπει ιδίω ε, να πρημοδοτήσουμε τους πιο φτωχούς πολίτες, τους άνεργους, τους άστεγους, τους φοιτητές και ο κύριος Χολμάγερ μας είπε ότι πρέπει να απευθυνθούμε ιδίω εις τους πιο φτωχούς πολίτες. Επίσης ε, προτείνει να απορρίψουμε ορισμένα τμήματα των τροπολογιών ε, και να μην υπάρξουν άλλες. Και τρίτον, ε, λέγει ότι δεν μπορούμε ε, να δεχθούμε μία απόρριψη ανοίγματο λογαριασμού. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τους λόγους. Βέβαια, το να προκαλέσει κανείς συλλογικές οικονομικές προσφυγές είναι υπερβολικό και δεν πρέπει εδώ να αναφέρονται. Ε, βλέπω ότι αναφέρει μάλιστα διάφορες συνμίσεις που δεν ξέρω τι είναι. Βοντεέρ, αντεέρ, έρελ, τι σημαίνει ε, εννοεί με το ΕΡ ριχτλίνια δηλαδή οδηγία ε, δεν θέλουμε να προκαταλάβουμε τη συζήτηση αλλά συλλογική συλλογική προσφυγή δεν πρέπει να επιτρέπεται διότι οι αποφάσεις θα πρέπει να κρίνονται κατά περίπτωση και οι τροπολογίες μέχρι και την δέκατη συμβιβαστική γίνονται αποδεκτές από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Έγγελ, ευχαριστώ και για τις μεταφράσεις τις οποίες μου προτείνατε. Φαντάζομαι ότι δεν έχουμε δυσκολίες να προχωρήσουμε και τώρα δίνω τον λόγο στον Όλε Σμιτ για τους φιλελεύθερους. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να ε, μιλήσω εξ ονόματός μου και αυτό είναι περίπλοκο, ξέρετε. Είναι πάρα πολύ καλή ε, η έκθεση που συντάξατε και σας το είπα το ίδιο απόγευμα όταν κάναμε τις συζητήσεις μας ε, και επί της ουσίας θα μπορούσα να συμφωνήσω με τις συμβαστικές ε, τροπολογίες. Κάναμε μια συζήτηση βεβαίως ε, για το επαχθές της διαδικασίας για τις τράπεζες. Ε, δηλαδή, τι είδους ε, με χρηματοπιστωτικούς κινδύνους θα διατρέξουν οι τράπεζες αν εφαρμοστεί αυτή η οδηγία. Και ένα από τα βασικά στοιχεία της τοποθέτησής μου είναι ακριβώς αυτό, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι αμφιλεγόμενο αυτό το ζήτημα, το ξέρουμε όλοι. Το να έχει κάποιο ένα βασικό τραπεζικό λογαριασμό, αν θεωρηθεί ότι συνιστά δικαίωμα για του καταναλωτέ, και θέλουμε έτσι να σχεδιάσουμε την εσωτερική αγορά, αν το πιστεύουμε αυτό, θα πρέπει να ε, φροντίσουμε ώστε να έχουν όλοι τη δυνατότητα να ανοίξουν ένα τέτοιο τραπεζικό λογαριασμό. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε πρόσθετα κολλήματα για όσους το επιθυμούν. Θα έλεγα ότι είναι κρίμα που τα κράτη-μέλη έχουν κάνει τόσα λίγα ώστε να δώσουν αυτά τα απαραίτητα εργαλεία στους ε, πολίτες τους. Αν βρούμε κάποιο κείμενο από το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε, κατά τη γνώμη μου, το βασικότερο ζήτημα είναι αυτό που λέμε στα γερμανικά ε, λογικό και κατάλληλο. ενώ το όφελος να είναι ε, αντίστοιχο του κόστους και του άχθους που συνεπάγεται το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού. Νομίζω ότι αυτό είπατε και θα μπορούσαμε ε, να συμφωνήσουμε. Νομίζω ο κύριος Χολμάγερ μέσω του συναδέλφου ε, Έγγελ αυτό εννοούσε ε, Στη συζητήση με τις τράπεζες και τις ενός τραπεζικών ιδρυμάτων νομίζω αυτό προκύπτει ούτως ή άλλως. Ένα άλλο βασικό, πάλι κατά τη γνώμη μου, είναι Ποια αιτιολογία δίνεται και βάσει ποιων κριτηρίων ε, ανοίγεται ένα τέτοιο βασικό τραπεζικό λογαριασμό, διότι στι ε, συζητήσει ε, αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να τεκμηριωθεί, να στοιχειοθετηθεί σχέση με το κράτο όπου ανοίγεται ο τραπεζικό λογαριασμό. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι συζητήσιμο. και έκανα τις προτάσεις μου ακριβώς επειδή είναι αφιλεγόμενο αυτό το ζήτημα. Ξαναλέω, πρώτον, είναι θέμα που πρέπει να ρυθμίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Β, μήπως είναι θέμα των κρατών μελών. Είναι δυνατόν να ε, καταστεί αυτό υποχρεωτικό για τις τράπεζες, η παροχή αυτής της βασικής υπηρεσίας. Εγώ θα απαντούσα καταφατικά και στις δύο ερωτήσεις. Έχει αλλάξει ο κόσμος και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει αυτό. Αν τώρα τα κράτη-μέλη που στο παρελθόν δεν έκαναν τίποτα, ε, κάποια, η πλειοψηφία ελπίζω, ε, θα συμφωνήσει να κινηθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν ξέρω, συνάδελφος πίσω που μας βάζει και τις ετικέτες, τι είναι αυτό τώρα φιλελεύθερο, σοσιαλιστικό, αυτό που λέω, γιατί τα είχαμε μπερδέψει όλα χτες ε, σε μια άλλη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι είναι δίκαιο για όλου. Ε, και είναι καλή συμφωνία και μπορούμε να το αποδώσουμε και στι προτάσει του κύριου Μόντι. Ε, με αυτόν τον τρόπο επαναδρομολογούμε την ε, εσωτερική αγορά και ικανοποιούμε έτσι ένα από τα αιτήματα του κύριου Μόντι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σμιτ. <clears throat> Δίνω τώρα τον λόγο ο κύριος Τούρνεν δεν είναι εδώ για τους πρασίνους και δίνω το λόγο στον κύριο Ντεζοντρίς για την ε, αριστερά. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ε, νομίζω ότι θα τον μπερδέψω ακόμη περισσότερο τον κύριο Σμίτε αλλά πάντως θα συμφωνήσουμε Ε, προτιθέμεθα να δεχθούμε κάποιες συμβαστικές ε, τροπολογίες ε, που μας φαίνονται θετικές. Η Γκουε θα μπορούσε να δώσει τη συγκατάθεσή της για αυτά τα βασικά ζητήματα. Για αυτό τον όρο reasonable, λογική σύνδεση, νομίζω ότι αναφέρθηκε ότι δεν θα πρέπει να μιλάμε παρά για το πραγματικό κόστος που συνεπάγεται το άνοιγμα ενός βασικού τραπεζικού λογαριασμού. Αν ναι, δεν το προσδιορίσουμε εμεί, ο καθένας θα μπορεί να ερμηνεύσει τον όρο reasonable. Νομίζω ότι όντω ε, θα ε, ήταν προτιμότερο να εξηγήσουμε, να προσθέσουμε αυτή τη διατύπωση που προτείνεται. Επίσης πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτή η σχέση με το κράτος Πώ θα αποδειχθεί. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε όλε τι καταστάσει οι οποίε θα χρειαζόταν κάποιο τραπεζικό λογαριασμό σε μια χώρα με του σκιώδει. Είπαμε παραδείγματο χάρη ε, ότι έχετε ένα τρίμηνο για να βρείτε μια θέση απασχόληση σε ένα κράτο μέλο. Αν δεν τα καταφέρετε, τι γίνεται. Αν έχετε πάλι οικογένεια σε κάποιο συγγενή σε κάποιο ε, κράτος μέλος ε, και κάποιο αποβιώνει, δεν θα ήταν ε, χρήσιμο να έχει κάποιο τραπεζικό λογαριασμό λόγω της έλλειψης εναρμόνιση του τραπεζικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ έχω τραπεζικό λογαριασμό στην Ολλανδία δεν σημαίνει ότι για οποιαδήποτε στιγμή μπορώ να κάνω οποιαδήποτε συναλλαγή η οδηποτε κράτο μέλο. Δεν υπάρχει αυτή, αυτή η ελευθερία. Όταν συζητάμε για μια σχέση με το κράτος. Ε, έχω να πω ότι δεν είναι εύκολο να ε, στοιχειοθετηθεί. Αυτό που μας μετέφερε ο κύριος Χολμαϊερ για το ODR-ADR επειδή μας έχει αποσχολήσει ε, αυτό το ζήτημα στην Επιτροπή μας, πιστεύω ότι είναι δύσκολο να ενσωματώσουμε και αυτό το στοιχείο μέσα στην έκθεση. Όταν ε, μια τράπεζα αρνείται να ανοίξει ένα τραπεζικό λογαριασμό, θα πρέπει να προβλέπετε ένα ένδικο μέσο, ένα τρόπο ε, προσφυγή ε, για τον πελάτη. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε και αυτό μέσα στην έκθεση. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να αναφερθούμε στο ADR ή στο ODR. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα. Πάντως ε, μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξή μας. Ε, e ευχαριστώ, Ντένις. Βλέπω ότι δεν είναι εδώ η ECR, αλλά βλέπω τώρα τον εκπρόσωπό τους και του δίνω το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εκ μέρους του κυρίου Φόρξ θα μιλήσω. Δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι παρόν σήμερα και ζητά συγγνώμη για την απουσία του ώστε να μπορέσει ο ίδιος ε, να εκφράσει τη θέση του. Λοιπόν, εγώ θα διατυπώσω τη δική του θέση όπως μου τη διαβίβασε. Η ομάδα ECR θα ήθελε περισσότερη προστασία για τον καταναλωτή. Είμαστε λοιπόν και εμείς της γνώμη ότι η πρόσβαση σε έναν βασικό τραπεζικό λογαριασμό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όμω, αυτή η νομοθετική πρόταση δεν είναι ο καλύτερο τρόπο για να επιτύχουμε τον επιθυμητό στόχο. Θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να επιτύχουν αυτό το στόχο σε εθνικό επίπεδο και αυτό αποδεικνύεται με τις εθελοντικές συμφωνίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με τις ε, τράπεζες για, την, για το άνοιγμα τέτοιων βασικών τραπεζικών λογαριασμών. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει την διερεύνηση όλων των δυνατών επιλογών πριν προβεί σε τελική νομοθετική πρόταση, έχοντας λάβει υπόψη πλήρως και την αρχή της επικουρικότητας. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Δεύτερο σχόλιο. Είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να έχουν επαρκή ευελιξία ώστε να εφαρμόσουν την πρόσβαση σε βασικέ τραπεζικέ υπηρεσίε. Γι' αυτό ασπαζόμεθα πλήρω την τροπολογία 41 τη κυρία Γκέπχαρτ. Δεν θα θέλαμε να είμαστε υπερβολικά περιοριστικοί για τον καθορισμό των όρων, ε, όπως τα κρατικά του λογαριασμού και η τιμολόγηση, ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν την επαρκή διακριτική ευχέρεια, ώστε να προσαρμοστούν στη δική τους τοπική αγορά. Θα μπορούσαμε να δεχτούμε και τη συμβαστική τροπολογία τη κ. Γκέπχαρτ, όπω υποβλήθηκε αυτήν την εβδομάδα ώστε αυτοί οι τραπεζικοί λογαριασμοί όσο το δυνατόν να είναι χωρίς χρεώσεις. Έπειτα, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσφοράς σε λογαριασμών από διαφόρους παρόχους, θέτοντας και, μάλλον η, α, η, θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων και υποχρεώσεων στους τραπεζικές ε, ιδρύματα δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Έπειτα, για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών θα πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ότι ταυτόχρονα με αυτό το δικαίωμα θα πρέπει να υπάρχουν και σχετικές διατάξεις ε, για την αντιμετώπιση της απάτης και του ξεοπλήματος βρώμικου χρήματος. Έπειτα, είναι λακτικέ όπως είναι η χρήση τραπεζικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου ή πιστοδικές κάρτες. Θα μπορούσαν λοιπόν αυτά τα μέσα να δώσουν τα ίδια αποτελέσματα, όπως είναι να καταδεθεί ένας ε, ε, μισθός κτλ. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι τα δικά μου λόγια, δεν είναι η δική μου θέση, είναι του κ. Φόξ. Αν έχω καταλάβει καλά τη θέση του, την οποία επαναλαμβάνω απλά, είναι έτοιμος ε, να δεχτεί είδη συμβασμού συνολικά το κείμενό σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Ευδία, ο κύριος Σαλβίνη απουσιάζει. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος, όχι. Ε, άλλοι ευρωβουλευτές, ε, μέλη της Επιτροπής. Θέλει κάποιος να παρέμβει πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι. Οπότε θέλω να, να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εάν θέλει να παρέμβει. Θα είμαι πολύ σύντομος, ε, κυρία Πρόεδρε. Είμαστε ευγνώμονε στην Επιτροπή σας, σε εσά προσωπικά και στους κοιόδης για αυτή την πρωτοβουλία. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, προσβλέπουμε ε, στην υιοθέτηση της ε, έκθεσής σας για να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Αν καταλαβα καλά, η ψηφοφορία θα γίνει αρχέ Ιουλίου ή τέλη Ιουνίου. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την τελική σας ε, έκθεση. vielen Dank. Ähm, Ευχαριστώ τότε σαν εισηγήτρια θα κάνω ακόμη μερικά σχόλια. Όντως, ε, θέλουμε τον Ιούλιο να θέσουμε το θέμα προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Βέβαια εξαρτάται από το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής και εμείς θα ψηφίσουμε ε, το 8 Μαΐου και ελπίζω ότι πολλά από τα πράγματα τα οποία θα συμφωνήσουμε θα υιοθετηθούν και ε, πρέπει να έχουμε μία συνεκτική πρόταση αλλά προτού αναφερθώ στο χρονοδιάγραμμα θα ήθελα να σχολιάσω ορισμένα θέματα που έθεσαν οι συνάδελφοι σχετικά με την αναγκαιότητα μίας νομοθεσίας επί του θέματος επί του οποίου υπάρχει ευρεία συνένεση στην Επιτροπή αυτή διότι είδαμε ότι παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από πέραν του ενός έτους ζήτησε από τα κράτη-μέλη να κινητοποιηθούν δεν έγινε τίποτα απολύτως στα κράτη-μέλη και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δεχθούμε έτσι δώσαμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να κινητοποιηθούν και γι' αυτό εμείς από ευρωπαϊκή σκοπιά πρέπει να κινητοποιηθούμε τώρα για να μπορέσουμε να θέσουμε τα θέματα σε κίνηση και συζήτηση. Όπως σας το πρότεινα θα ήθελα να παραμείνουμε στο συμβιβασμό που προτείνω και να μιλάμε για τα όσο το δυνατόν λιγότερο κόστος ή με αντίστοιχο κόστος γιατί όπως είχα πει ή στην συζήτηση ε, στους συντονιστές θεωρώ προβληματικό να θέσουμε ένα ανώτατο επίπεδο 5 ευρώ ή 12 ευρώ διότι υπάρχει διαφορετικό βιωτικό επίπεδο στα διάφορα κράτη. Και για τη Γερμανία 5 ευρώ δεν είναι πολύ, ενώ μπορεί για τους Ρουμάνους να είναι ένα τεράστιο ποσό. Ως εκ τούτου δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να προχωρήσουμε έτσι και απλώς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το επίπεδο τιμών στα κράτη-μέλη και αυτό είναι η πιο λογική διατύπωση και παραμένω στην πρότασή μου. Όσο αναφορά περαιτέρω άλλα σχολεία. Προσπαθώ να συμφωνήσω με το ΕΛΚ και θέλω να πω σαφώς ότι δεν μπορεί κανείς ε, να, να ζητήσει μία αποδεδειγμένη σύνδεση διότι δεν έχουμε ε, ε, καμία απόδειξη αν κάποιος δεν έχει μία διεύθυνση και έναν λογαριασμό σε ένα κράτος αλλά σέβομαι τα παραδείγματα που ανέφερε ο Ντένις, δηλαδή εάν βρίσκουμε σε μία χώρα, σε διακοπές και θέλω να ανοίξω ένα λογαριασμό για τα γενικά μου έξοδα ή σαν φοιτητή να επαρκεί ε, να πούμε ότι έχω αυτό το λογαριασμό στο διαδίκτυο και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ε, έχω λύσει με τις προτάσεις μου για το collective regret ε, είναι μία έννοια η οποία απλώς επαναλαμβάνει την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν το προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγώ γιατί να το απορρίψω. Απλώς στηρίζω αυτά τα οποία έπραξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του θέματος, αν και στην διατύπωση δεν υπάρχει προϋπόθεση ε, η οποία προκαταλαμβάνει τι θα κάνουμε στην νομοθεσία που θα προτείνουμε και γι' αυτό υπάρχει και η τροπολογία γιατί όντως οι κανόνες τους οποίους εμείς καταρτίζουμε θα πρέπει να διευκρινιστούν κατά περίπτωση. Όσον αφορά το mobile banking προς τον κύριο Έγγελ θέλω να διευκρινίσω στην Ρουμανία και στη Βουλγαρία γιατί υπάρχουν τόσοι που δεν έχουν είναι λογαριασμό γιατί σε ορισμένες περιοχές δεν υπάρχουν τράπεζες. Πρέπει λοιπόν κανείς να έχει πρόσβαση στο λογαριασμό του και γι' αυτό μπορεί να επιλέξει, να επιλέξει το web banking. Ε, δεν ε, συνεπάγεται μεγάλα έξοδα και για να αποφύγουμε ε, να μεγαλώνουν τα έξοδα θα πρέπει να κοιτάξουμε στα κράτη με ωφέλη, ποιες είναι οι λύσει οι οποίες μπορεί να είναι κατάλληλε και νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή το web banking είναι η κατάλληλη λύση και γι' αυτό το προτείνω διότι στην εκ πρώτης όψεω ίσως δεν είναι προφανές αυτά είχα να σας πω στα διάφορα θέματα που αναφέρθηκαν και θα δούμε στη συνέχεια πόσο θα προχωρήσουμε. Εγώ είμαι επιφυλακτική, ελπίζω όμως ότι θα έχουμε στο τέλος καλές συμβιβαστικές τροπολογίες. Αυτό απέδειξε και η συζήτηση σήμερα και σας υπενθυμίζω ότι στην Επιτροπή θα ψηφίσουμε στις 8 Μαΐου και υπενθυμίζω στους κοιόδης εισηγητές ότι περιμένω τα σχόλια στο κείμενό μου μέχρι αύριο το μεσημέρι για να μπορέσω να το επεξεργαστώ περαιτέρω και στη συνέχεια να διατυπώσω τα κείμενα που μπορώ να σας αποστείλω εγκαίρως. Όσον αφορά την Οικονομική Επιτροπή, η ψηφοφορία θα είναι στις 31 Μαΐου και ελπίζουμε ότι θα μπει στην ημερήσια διάταξη του Ιουλίου για την Ολομέλεια. Μετά την προεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αυτή τη στιγμή σκέφτεται πώς πρέπει να προχωρήσει. Σας επιθυμίζω άλλωστε ότι πρόκειται για μία νομοθεσία θετική πρόταση κατά πρωτοβουλία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συμπεριφερθεί αναλόγως, ιδίως για ένα τόσο σοβαρό θέμα που μας απασχολεί όλους. Εάν δεν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να παρέμβει, μπορώ να κλείσω τη συζήτηση στο θέμα αυτού και προχωρώ στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο κύριος Μπουσουτήλ είναι εδώ, το Internal Market scoreboard ε, πίνακας ε, αποτελεσμάτων εσωτερικής αγοράς. Κύριε Μπουσουτήλ, προσέξτε με γιατί απευθύνομαι σε εσά για τη δικιά σας έκθεση. Ε, τον πίνακα αποτελεσμάτων εσωτερικής αγοράς. Στις 10 ε, παρατέταρτο προβλέπεται η ψηφοφορία. Έχουμε ακόμη τρία λεπτά και θα περιμένω ακόμη τρία λεπτά πριν ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες αλλά εσείς ε, κύριε Μπουσουτήλ θα μπορούσατε να υποφιληθείτε να σχολιάσετε εντωμεταξύ το κείμενό σας. Εάν θέλετε σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω μαλτέζικα. Διότι ο Φρανκ που είναι δίπλα μου μου είπα θέλει να ακούσει πώς ακούγονται δηλαδή τα μαλτέζικα. Γιατί του φαίνονται πολύ πιο ενδιαφέροντα τα μαλτέζικα από τα γερμανικά. Υπάρχουν 66 τροπολογίες, ε, η μία έχει αποσυρθεί. Και έχουμε τέσσερις συμβαστικές τροπολογίες. Θα ήθελα να σας ενημερώσω, Πρόεδρε, ότι θα καταθέσουμε και δύο προφορικές τροπολογίες. Η μία από τον υποφαινόμενο και αναφέρεται στην τροπολογία 38 αυτή η προφορική τροπολογία. Ο κύριος Κάρας θα καταθέσει άλλη μία προφορική τροπολογία. Με ακούτε, με παρακολουθείτε. Μάλιστα κυρία Μπουσούτιλ, σας παρακολουθούμε. Μπορείτε να συνεχίσετε. Okay, orali. Έχουμε δύο προφορικές τροπολογίες, έλεγα λοιπόν. Η μία είναι δική μου και αναφέρεται στην τροπολογία 38 και η άλλη του κυρίου Ότμαν Κάρας και αναφέρεται στην 18β. Ε, κατόπιν τούτων μπορούμε να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πάντως τους Κιώδης για τη βοήθεια τους. Χάρη σε αυτήν ε, βελτίωσα την έκθεση μου σε σχέση με το πρώτο σχέδιο που είχα καταθέσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπουσουτήλ. Ε, εκπρόσωπος ε, των σοσιαλιστών. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να επισημάνω πόσο καλή ήταν η ατμόσφαιρα στις διαπραγματεύσεις που μας οδήγησαν σε αυτή την έκθεση. Αλλά ταυτόχρονα θέλω να εκφράσω και μία λύπη. Γιατί δεν μπορέσαμε να να περάσουμε την τροπολογία την προφορική τροπολογία, καθώς είναι περίπλοκο νομικό ζήτημα που υπευλήθη χθες. Μόλι χθε και δεν είχαμε τότε να μελετήσουμε εις την αυτροπολογία. Τρέφω λοιπόν σοβαρέ αμφιβολίε. Και πώς γίνεται δηλαδή πέντε μήνε μετά από τόσο επικοδομητική συζήτηση προκύπτει μια τέτοια τροπολογία τόσο περιπλοκή που δημιουργεί πολλά νομικά ερωτηματικά. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλοι σκιώδεις εισηγητές που θα ήθελαν ακόμη να παρέμβουν. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι τέτοιο. Οπότε παρακαλώ να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία Κατόπιν αυτού, προτού ξεκινήσουμε την ψηφοφορία, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι μετά τις δύο ψηφοφορίες που θα έχουμε εδώ, θα υπάρξει και μία ψηφοφορία σχετικά με την πρόταση των συντονιστών εχθές το βράδυ για την έκθεση της κυρίας Κόμη, διότι οι συντονιστές προτείνουν να την ψηφίσουμε σε πρώτη ανάγνωση και αυτό πρέπει να τεθεί προς έγκριση στην Ολομέλεια με ε, την συνένεση 21 μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οπότε ε, μετά τις ψηφοφορίες μην φύγετε αμέσως η κυρία Ρούλε ε, δεν θα έλεγα οι συντονιστές θα έλεγα έλεγα η πλειοψηφία των συντονιστών διότι δεν ψηφίσαμε και εγώ εξέφρασα τις επιφυλάξεις μου. Ευχαριστώ. Όντως επαναλαμβάνω τη διατύπωση που χρησιμοποίησα σήμερα το πρωί δηλαδή ότι μετά από μακρά συζήτηση οι συντονιστές απεφάσισαν να προσπαθήσουν, να προσπαθήσουν δεν σας είπα ότι εσείς συμφωνήσατε επαναλαμβάνω αυτά που είπα σήμερα το πρωί. Ε, δηλαδή, αν με αφήσετε να τελειώσω τη φράση μου, ότι θέλουμε να κάνουμε μία προσπάθεια να περάσουμε το θέμα αυτό στην Ολομέλεια σε πρώτη ανάγνωση και αυτό ε, έτυχε τη συνένεση της πλειοψηφία των συντονιστών χωρίς να θέλω να συμπαρασύρω την κυρία Ρούλε η οποία σαφώς αντετέθη. Σωστά μου το είπατε και δεν, θέλω, δεν το υποτιμώ καθόλου. Κατόπιν λοιπόν αυτών των δύο ψηφοφοριών θα προβούμε σε αυτή την ψηφοφορία που προανέφερα. Τώρα προχωράμε στην έκθεση του κυρίου Μπουζουτήλ και αναφέρομαι καταρχήν στην τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά ερχόμαστε στην προφορική τροπολογία του κυρίου Μπουσουτήλ Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η προφορική τροπολογία είναι η εξής. Είναι η συνέχιση της τροπολογίας 38 η οποία στο τέλος θα προσθέτει. Ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσει μία διαδικασία ταχείας αντιμετωπίσεως των παραβιάσεων και να προβλέψει την κατάρτιση εσωτερικής αγοράς και του σχετικού δημοσίου κατηγορίου δικηγόρου ώστε να προετοιμάζεται η διαδικασία αυτή ανεξάρτητα από αυτές οι οποίες ε, ε, απαιτούν έγκριση από τους επιτρόπους. Κοιτάτε, αυτή η νέα προφή ενός ε, νέου εισαγγελέα, ενός prosecutor που θα παρακολουθεί αυτές τις διαδικασίες είναι κάτι πολύ περίπλοκο και σημαντικό και δεν μπορώ να δεχτώ μια τροπολογία μόλις 12 ώρες πριν ψηφοφορία. Στο ε, συγγνώμη. Ο κύριος Ντεζά. Ευχαριστώ. Ε, συμφωνώ και εγώ, διότι έχω έχει γίνει αυτή η συζήτηση και Νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει αυτό το θέμα και ξέρουμε τι περιέχει αυτό το έγγραφο, κυρίω σε σχέση με, αυτά, ε, με την αναφορά στον εισαγγελέα. Δεν μπορούμε όμως να ανοίξουμε καινούργια ζητήματα εδώ. Ε, λοιπόν, κύριε Άγγελε, εντάξει, αλλά τελευταίος παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επειδή καταρχήν ε, είχα τις ε, ίδιες επιφυλάξεις και συζήτησα με τον κύριο Μπουσουτήλ, μπορώ να σχολιάσω το εξής για, το, για πίσω τον κύριο Ντεκάμπους και τον, τους άλλους συνεδέρφους ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Μπορούμε να θέσουμε ε, ε αλλά αυτό δεν, δεν ισχύει για το κείμενο του Κοινοβουλίου. Μπορούμε όμως να μιλούμε εφόσον λέμε to consider establishing απλούστατα ε, μιλάμε ότι ε, το σκεφτόμαστε σκεφτόμαστε για να επιζητήσουμε ένα συγκεκριμένο ε, στόχο Παρακαλώ λοιπόν τον κύριο Ντε Γιόγκ να μην αντισταχθεί. Ε, ευχαριστώ κύριε Έγγελ. Δύο συνάδελφοι είναι κατά ε, και ε, κατόπιν αυτού δεν μπορεί να ψηφιστεί έτσι μία προφορική τροπολογία και μέχρι την Ολομέλεια μπορείτε να συζητήσετε και να δείτε αν θα κάνετε κάποια άλλη τροπολογία σε αυτήν. 38 υπέρ. Κατά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 κατά ε, παρακαλώ δεν πρέπει ήδη να κουραστήκατε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά έρχομαι στην παράγραφο 18 που υπάρχει η τροπολογία προφορικά του Ότμαρ Κάρας. Με συγχωρείτε, είναι μετά την τροπολογία 56, οπότε 55 ε, τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η κυρία Χάνσλικ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Κάρος μου ζήτησε να διαβάσω μια προφορική τροπολογία για το άρθρο 18β. Να το διαβάσω στα αγγλικά ότι επιβεβαιώνουμε τη συμμετοχή των συνδεμένων εταίρων στα πλαίσια του Solvit, ιδίως με στόχο την αύλυνση του ιδιαίτερου βάρους και επισημαίνει ότι η συνεργασία με τους εταίρους έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στον παρελθόν μεταξύ άλλων λόγω της άμεσης επαφής ε, με τους πολίτες. Καλή, λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η πρόσβαση των συνδεδεμένων εταίρων στο Solvit είναι κάτι που θα διατηρηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Χάνσλι. Υπάρχουν παρεμβάσεις από αυτού, Αντώνιο, όχι. Τότε μπορούμε έτσι να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμφωνείτε αν ψηφίσουμε από κοινού την 63, 64, 65, ναι, ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνονται. Και τώρα ερχόμαστε στην τροπολογία 1, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ και 4 και 5 μάλλον όλες μαζί συμφωνείτε υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 και 9 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται Δέκα. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αυτό πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος Τροπολογία 11. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Ο κύριος Μπουσουτήλ δεν έχει την κάρτα του, οπότε ε, μήπως κάποιος άλλος ξέχασε την ε, κάρτα του. Ε, τότε κλείνω την ψηφοφορία. Τώρα έκλεισα την ψηφοφορία και έχουμε 19 ε, υπέρ, 11 κατά, άρα αποδεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 14 απεσύρθη, η 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού από τη 18 μέχρι την 23 ευχαριστώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το ψήφισμα όπως έχει τροποποιηθεί ε, ψηφίζεται ηλεκτρονικά, ξεκινάει η ψηφοφορία. Κύριε Μπουσουτήλ θα σας συνυπολογίσουμε στους υπέρ, οπότε ε, κρίνουμε την ψηφοφορία και έχουμε 31 υπέρ καμία αρνητική ψήφος, καμία αποχή. Σας συγχαίρω για το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Και τώρα ερχόμαστε στην ε, ε, ψηφοφορία της εκθέσεως της Μαρία Ιριγκοένε Περές σχετικά ε, με τους καταναλωτές. Θέλεις το λόγο για λίγα λεπτά, Μαρία. Για ένα λεπτό. Όχι Είναι. Καλημέρα σας και ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ όλες τις πολιτικές ομάδες για την συνεργασία τους για να εκπονήσουμε αυτή την έκθεση για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών, ώστε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά στην ολοκλήρωση της ιστορικής αγοράς. Ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία. Ευχαριστώ. Μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία εάν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια από τους χειώδεις εισηγητής που δεν βλέπω. Συμβιβαστική 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβιβαστική 14. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ η 35 Αντώνιο 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά νομίζω ότι εδώ θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά σχετικά με την τροπολογία 61 τρο... ηλεκτρονικός έλεγχος ξεκινάει η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι λίγοι 13 υπέρ 15 κατά απορρίπτεται δηλαδή και αυτό λύνει το πρόβλημα και για την 60 58 ε, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 σαν προστίκι υπέρ κατά αποχή εγκρίνεται 57. Επίσης σαν προσθήκη υπέρ. Αλλά πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. 13 υπέρ, 16 ε, κατά, άρα απορρίπτεται. Τροπολογία 63 υπέρ. Και πάλι ηλεκτρονικός έλεγχος, ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία. Τώρα, τώρα μάλλον. 15 υπέρ, 13 κατά. Δηλαδή ε, εγκρίνεται η τροπολογία 63 ε, σαν προσθήκη 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και έτσι καταπίπτουν όλες οι επόμενες τροπολογίες διότι διαγράφονται συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά και εδώ θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση ξεκινάει τώρα ψηφίσατε όλοι λίγη ψηφοφορία 15 υπέρ 12 κατά άρα εγκρίνεται η 84 σαν προσθήκη υπέρ Επίσης ηλεκτρονικός έλεγχος ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. 16 υπέρ 13 κατά. Εγκρίνεται. 83 σαν προσθήκη. Ποιος είναι υπέρ. Και εδώ ηλεκτρονικός έλεγχος ξεκινάει. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. 18 υπέρ 10 κατά και εγκρίνεται. Τροπολογία 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, κατά αυτόν τον τρόπο καλύπτεται και 36, 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ εδώ ψηφίζουμε ηλεκτρονικά ξεκινάει η ψηφοφορία σχετικά με την 88 ψηφίσατε όλοι λίγοι 16 υπέρ 13 κατά η συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ ηλεκτρονική επαλήθευση ξεκινάει. Ψηφίσατε όλοι, λίγοι, 17 υπέρ, 12 κατά και εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Με συγχωρείτε, ξέχασα την τροπολογία 98 που προηγεί το της 107 σαν προσθήκη στην συμβιβαστική 9 και μπορεί να ψηφιστεί. Παρακαλώ λοιπόν, σχετικά με την 98, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Ερχόμαστε τώρα στην 108, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 ηλεκτρονικός έλεγχος ξεκινάει η ψηφοφορία ψηφίσατε κλείνει 13 ε, υπέρ 16 κατά απορρίπτεται λοιπόν η 111 ήταν αυτή λοιπόν η 110 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 ηλεκτρονική επαλήθευση ψηφίσατε λίγοι 13 υπέρ 16 κατά η 126 σαν προσθήκη ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ ηλεκτρονική επαλήθευση ξεκινά ψηφίσατε όλοι λίγοι 30 ναι, 16 ε, όχι. 13 ναι και 16 όχι. 133 υπέρ, κατά. Επανέρχομαι. Συμβιβαστική 13, γιατί σιγά σιγά κουράζεστε. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Ξεκινάει. Ψήφισαν όλοι. Λίγοι. 18 υπέρ 11 κατά. Εγκρίνεται. 146. μάλλον ε, δεν ε, ισχύει πλέον και πάμε στην 143 διότι και 144 καταπίπτει για την 143 ποιος είναι υπέρ ηλεκτρονική επαλήθευση ξεκινά ψηφίσατε λίγοι 13 υπέρ 15 κατά απορρίπτεται 142 ηλεκτρονικά Ξεκινά. Λίγοι. 12 υπέρ, 16 κατά, απορρίπτεται. Ε, 34 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. 15 υπέρ 12 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Επίσης ηλεκτρονικά. Ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Ε, κλείνει 13 υπέρ 16 κατά. Ε, τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασ... Ε, τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15, ε, τροπολογία 10, σαν προσθήκη, ε, για να προσθήσουμε τον όρο gender. Ποιος είναι υπέρ. Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Λίγη ψηφοφορία. 14 υπέρ, 13 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το ψήφισμα όπως τροποποιήθηκε. Ε, ποιος είναι υπέρ ηλεκτρονικά. Με συγχωρείτε, πρέπει να γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση για να καταγραφεί το αποτέλεσμα, οπότε ηλεκτρονική ψηφοφορία, αν ψηφίσατε όλοι, κλείνει η ψηφοφορία. 28 υπέρ, ένας κατά, καμία αποχή. Κυρία Ερυγκογέν Περές, σας συγχαίρω για την καλή εργασία και το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, τώρα έχουμε άλλη μία ψηφοφορία η οποία αναφέρεται στην πρόταση των συντονιστών σχετικά Παρακαλώ να είστε λίγο ήρεμοι για να ακούγομαι σχετικά με τη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση για τις διαπραγματεύσεις της εκθέσεως ε, της κυρίας Κόμη. Πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά. Παρακαλώ λοιπόν να ξεκινήσει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Λίγοι. 25 υπέρ και 3 αποχές. Οπότε έτσι απεφάσισε η Επιτροπή ότι θα προχωρήσουμε στη συζήτηση σε πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε τις ψηφοφορίες και θα δώσω τον λόγο και την... Ε, θα δώσω τον λόγο αλλά όχι την Προεδρία στην Μπάρμπαρα... και την Προεδρία στην Μπάρμπαρα Βάιλερ και σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. C'est très important pour une commission. Oui. Mm.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 παρακαλώ τους συναδέλφους και τους σκιώδεις ε, τους οποίους βλέπω εδώ βλέπω ότι δεν είναι εδώ όλοι οι σκιώδεις και παρακαλώ να προσέλθουν Ωραία. Ας ε, συνεχίσουμε. Ε, ελπίζω ότι θα έρθει και νωρίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα τρία τελευταία θέματα της μερισίας διατάξεως για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα και τώρα θα συζητήσουμε την επόμενη εκθεσή και δίνω το λόγο στην κυρία Βάισμπεργκερ για την ηχοστάθμη των μηχανοκινήτων οχημάτων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είναι ένας περαιτέρω φάκελος ο οποίος ασχολείται με τα αυτοκίνητα και εδώ δεν πρόκειται για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά με την ηχορύπανση και για τα αυτοκίνητα δηλαδή να μην κάνουν τόσο θόρυβο τα ιδιωτικά οχήματα και τα οχήματα δημοσίας χρήσεως διότι ο συνεχής θόρυβας μπορεί πέραν των ασθενειών να προκαλέσει διαταραχές του ύπνου και άλλες και έχουμε 2.010 ε, εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι υφίστανται ε, πολύ υψηλή χορύπανση. Άρα πρέπει να προστατεύσουμε την ε, ποιότητα ζωής των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την υγεία τους. Και μειώνει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, το επίπεδο των ε, ήχων ε, και της ηχορύπανσης σε χαμηλότερα επίπεδα, δηλαδή έχει περιλάβει όλα τα οχήματα και τα μειώνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ξεκινά σε δύο χρόνια, η δεύτερη μετά από πέντε χρόνια, δηλαδή όπως βλέπετε είναι ασφιχτική εκρηκτικές ε, οι προθεσμίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έτσι η επιβάρυνση της συγχωρηπάνσεως μειώνεται κατά 25% σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά θέλουμε να υπάρχει και ένα νέο μηχάνημα μετρήσεως της συγχωρηπάνσεως ε, και ο έλεγχος αυτός ε, θα μπορέσει να προσαρμοστεί στην συγκοινωνία της πόλεως που έχουμε λιγότερο λιγότερες επιταχύνσεις και περισσότερες, ε, και περισσότερες φορές ξεκίνημα σταμάτημα. Είναι λοιπόν μία πολύ μακριά διαδικασία για να προσαρμοστούμε σε, αυτές, ε, σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Θέλω να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος η οποία ηγείται επί του θέματος έχει θέσει ένα πολύ στενό χρονικό περιθώριο μέχρι μέχρι τις 10 Ιουλίου για ψήφιση και εγώ ζήτησα εγκαίρως να κάνουμε γνωμοδότηση, άργησε να ληφθεί η απόφαση και τώρα πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Γι' αυτό και την περασμένη εβδομάδα έδωσα το έγγραφό μου προς μετάφραση και ε, θα το υποβάλω σήμερα το απόγευμα γραπτός εις ε, τους ε, στους μεταφραστές και προσπαθώ να δω πώς ε, θα μπορέσει η γνωμοδότηση αυτή από πλευράς των καταναλωτών ε, να προσαρμοστεί. Καταρχήν με ενδιαφέρει η ενημέρωση των καταναλωτών. Αυτό είναι και ο στόχος μας να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια για τους καταναλωτές σχετικά με τις πληροφορίες. Ε, προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η Επιτροπή μας. Έχουμε μία σήμανση, παραδείγματο χάρη, σχετικά με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος και ε, με τον θόρυβο των ελαστικών πάνω στις ρόδες. Σήμερα όμως δεν έχουμε ε, πρότυπα για τις εκπομπές θορύβου και θα πρέπει να ενημερώνουμε τους καταναλωτούς με μία συγκρίσιμη και σαφή σήμανση πράγμα το οποίο ισχύει και για όλα τα άλλα στοιχεία όσον αφορά τα άλλα θέματα της εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος όπου δεν λέγονται οι οριακές τιμές που προτείνονται ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσει έναν κανονισμό για την σήμανση και να δούμε τι πρέπει να γίνει ε, και πώς μπορούμε να προτείνουμε στη σήμανση σήμανση για το διοξίδιο του άνθρακος και μία σήμανση για το θόρυβο. Γιατί, διότι παραδείγματο χάρη για την ε, ε, τα οχήματα δημοσίας χρήσεως υπάρχουν προβλήματα σε ορισμένες ε, κοινότητες όπως στην Ολλανδία λέγεται ότι τα φορτηγά που παραδίδουν τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ δεν πρέπει να ξεπερνούν ένα επίπεδο θορύβου. Υπάρχουν δηλαδή προδιαγραφές ε, για αυτή την ηχορύπανση και πρέπει να δούμε ε, τι γίνεται τελικά διότι ε, ούτως ή άλλως υπάρχουν ορισμένα μέτρα τα, μέσα τα οποία αγοράζονται ακριβώς για να είναι θορυβόδη αλλά θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του και την περαιτέρω χρήση. Ένα άλλο θέμα για μένα είναι ότι θέλουμε να υπάρξει ένας μακροπρόθεσμος στόχος, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως σας είπα, προτείνει δύο φάσεις, δύο χρόνια και μετά άλλα τρία σύνολο πέντε, που κατά τη γνώμη μου δεν είναι επαρκή. Πρέπει μακροπρόθεσμα να μειώσουμε και περαιτέρω το θόλυβο, και έτσι θα βελτιώσουμε την προστασία της υγείας των καταναλωτών με τη μείωση του θορύβου, θα υπάρχει νομική ασφάλεια και σαφή στοιχεία για τους, καταναλωτε... για τους κατασκευαστές, να ξέρουν δηλαδή ε, τι μπορούν να προτείνουν και ε, πρέπει αυτά να συμπληρωθούν και ε, πρέπει να προτείνουμε μακροπρόθεσμο στόχο κατά τρόπον ώστε να ξέρουμε πού θα καταλήξουμε ε, ο δεύτερος λοιπόν στόχος είναι μακροπρόθεσμη ρύθμιση. Τρίτον, να υπάρχει μία διαφοροποίηση μεταξύ ε, των φορτηγών και των οριακών τιμών, διότι υπάρχουν ε, κατηγορίες οχημάτων και υπάρχουν οριακές τιμές στο παράρτημα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατακρίνεται γιατί το παράρτημα αυτό οι κατηγορίες ε, των οχημάτων δεν ξεχωρίζουν επαρκώς. Εγώ λοιπόν προτείνω τέσσερις κατηγορίες ε, στις διάφορες κατηγορίες ε, προβαίνω σε μία διαφοροποίηση κατά τρόπον ώστε να προσαρμόζομαστε στο είδος του οχήματος και να υπάρχει μία δίκαιη και ρεαλιστική προσπάθεια μειώσεως του θορύβου. Κοίταξα λοιπόν το τον κατάλογο αυτό συζήτησα με τους ενδιαφερόμενους την βιομηχανία, τους οδηγούς και υπάρχει μία νέα πρόταση με τη διαφοροποίηση απλή η οποία βασίζεται στη γνώμη των εμπειρογνωμόνων και αν κοιτάξουμε ε, το κατάλογο αυτό θα δείτε μία περαιτέρω πρωτότυπη ιδέα μου που διαχωρίζει τα ιδιωτικά οχήματα από τα οχήματα δημοσίας χρήσεως διότι ο κύκλος ζωής είναι διαφορετικός στις δύο περιπτώσεις ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει το ίδιο χρονικό περιθώριο και για τις δύο κατηγορίες ενώ νομίζω ότι θα πρέπει να διαχωρίσει κανείς από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα από τα δημοσία χρήσεως. Επίσης πρέπει να δούμε τα θέματα από την πλευρά του καταναλωτή, δηλαδή δηλαδή πώς οι οριακές τιμές αυτές μπορούν ε, να επηρεάσουν ε, το κόστος του αυτοκινήτου ε, πράγμα που μας οδηγεί να σκεφτούμε τι συνεπάγεται και θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ορισμένες τεχνολογίες οι οποίες μειώνουν το θόρυβο αλλά έχουν παρενέργειες αν δεν υπάρξει ένα νέος κινητήρας βλέπουμε ότι με την encapsulation ε, κλείνουμε τον κινητήρα σε ε, ένα περίβλημα και μπορεί κανείς να αυξήσει την θερμοκρασία και σε μία μακριά διαδρομή να υπερθερμανθεί ο κινητήρας. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις οριακές τιμές. Επίσης η ε, θόρυβη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων τον πράγμα το οποίο είχε μεγάλη επίχυση στα δημόσια μέσα ενημέρωση στη Γερμανία και για να διατυπώσω σωστά την πρόταση θέλω να πω ότι όντως υπάρχει κίνηση διότι ε, με μικρή ταχύτητα ο πεζός εάν είναι μεγάλη η, η ταχύτητα ακούγεται ο θόρυβος των ελαστικών αλλά στη μικρή ταχύτητα δεν υπάρχει υπάρχει κανένας θόρυβος και υπάρχει κίνδυνος για τους τυφλούς πεζούς. Δεν μπορώ να υποχρεώσω να υπάρξουν αυτοί οι θόρυβοι, αλλά αν οι κατασκευαστές αποφασίσουν να υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση του θορύβου στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα πρέπει να γίνει εναρμονισμένα και συντονισμένα. Δηλαδή, ε, έχουμε δει πρωτότυπες και αρνητικές προτάσεις ότι ε, δεν μπορούμε ε, τα αυτοκίνητα αυτά να έχουν τεχνητούς ήχους, δηλαδή ε, ήχους από ζώα. Είναι γελία πράγματα. Δεν μπορούμε εμείς να προδιαγράψουμε τι θόρυβος θα υπάρχει, απλούστατα να έχουν όλοι τον ίδιο θόρυβο. Και στο σημείο αυτό, κυρία Πρόεδρε, πρέπει να σας πω ότι είχαμε ζητήσει ενισχυμένη συνεργασία, διότι εδώ ασχολούμαστε με την προστασία σημασία της υγείας και στο σημείο αυτό εάν θέλω όντως να υπάρξουν θόρυβοι τότε ε, δεν, ε, δεν θα υπάρξει μία, ε, μία μονομερής ρύθμιση και ζητήσαμε όπως σας είπα την ενισχυμένη συνεργασία υπάρχει τώρα η προϋπόθεση από ό,τι γνωρίζω αλλά σχετικά με το άρθρο 50 δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την use procedure, να μην πάμε κατευθείαν στην Ολομέλεια, αλλά να ξαναγυρίσει η γνωμοδότησή μας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και εφόσον πρόκειται για προστασία των καταναλωτών και για εναρμόνιση, νομίζω ότι μπορούμε να κινηθούμε άμεσα και όχι μέσω της Επιτροπής Περιβάλλοντος. 8 ε, Μαΐου θα ξανασυζητήσουμε βάσει της γραπτής εκθέσεως και αυτό που ελπίζω είναι ότι θα έχουμε επαρκή χρόνο μέχρι τις 15 Μαΐου για τροπολογίες και ε, θα ήθελα να απευθυνθώ στους άλλους συντονιστές και να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κοινέ τροπολογίες οι οποίες θα συζητηθούν ψηφιστούν στις 20 Ιουνίου, θα ψηφιστούν στις 21 Ιουνίου και έχουμε καιρό μέχρι τις 10 Ιουλίου στην Ολομέλεια κατά τρόπον ώστε το σχέδιό μας να εσωματωθεί στο τελικό κείμενο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η εισαγωγή σας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ε, κυρία Βέστφαλ, με συγχωρείτε, προχωρήσαμε ήδη, αλλά εξοικονομήσαμε μισή ώρα από τις ε, ψηφοφορίες και μπορούμε τώρα να τις χρησιμοποιήσουμε. Ο κύριος Μάντερς όμως έχει εντωμεταξύ εγκαταλείψει την αίθουσα. Θα ξανάρθει, δεν ξέρετε. Λοιπόν, Επόμενη εισηγήτρια η κυρία Βέσφαλεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφε, ε, αγαπητή κυρία Δόκτωρ Βάις Γκέμπερ. Βέβαια δεν σημαίνει ότι το θέμα αυτό είναι λιγότερο ενδιαφέρον αλλά θα ήθελα να κάνω ορισμένε ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά φαντάζομαι ότι θα τις μεταβιβαστούν. Καταρχήν χαιρετίζουμε την πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεωρεί τον θόρυβο της κυκλοφορίας σαν ένα πεδίο μάχη, είμαι παλιά καραβάνα στην πολιτική και ξέρω ότι κάθε όχημα υπόκειται ένα τεστ θορύβου και είναι πολύ σημαντικό ιδίως για τους ανθρώπους που ζουν στις πόλεις και στις μικρές κοινότητες και υφίστανται τους θορύβους αυτούς και την ηχορύπανση. Ε, πρέπει να πω ότι η τωρινή πρόταση είναι πολύ πιο ρεαλιστική από το ισχύον σύστημα εξετάσεως που είναι πιο παλιό. Δεν άκουσα την εισαγωγή της κυρίας Βάις Γκέρμπερ, αλλά υποθέτω ότι θα υπάρξουν παρεμφερείς ερωτήσεις, αλλά ε, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να έχουμε α απαντήσει στα ερωτήματα και θα ήθελα να ρωτήσω εάν η πρόταση βασίζεται ή στις παλιές κατηγορίες οχημάτων και εμείς ακούμε από πολλούς τομείς ότι οι κατασκευαστές δεν αντέδρασαν. Δηλαδή ε, αυτό ε, προκαταλαμβάνει ε, την ασφάλεια ασφάλεια προγραμματισμού. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι λαμβάνονται υπόψη ε, οχήματα ε, τα οποία είναι πολύ παλιά και αντιπροσωπεύουν πλέον μόνο 5% των κυκλοφορούντων ε, ε, οχημάτων. Εάν όλα αυτά ισχύουν, τότε θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι η διαδικασία των δοκιμών ε, δεν θα αποδώσει. Και πέραν αυτού θα ήθελα να ξέρω τι προβλέπετε ε, με τις νέες τιμές, διότι άκουσα ότι ουσιαστικά εδώ αναφερόμαστε ιδίως στις κατηγορίες αυτοκινήτων μη 1, μη 2, νη 2, μη 3 που θα έπρεπε όμως ε, να ε, τεθούν σε χαμηλότερη μοίρα διότι ε, η μεγαλύτερη χορύπανση υπάρχει σε μεγάλες σε κατηγορίες μεγάλων οχημάτων και επιπλέον υπάρχουν και ορισμένες άλλες και αναρωτιέμαι εάν δεν υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αυτό όσον αφορά τις προτάσεις που έχω για τις τεχνικές προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η αξία της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πράσινη βίβλο του 1996 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε θεωρήσει ότι το 20% του πληθυσμού υπό βάλετε σε μια χορύπανση η οποία είναι αφόρητη και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εντοπίσει τις διάφορες πηγές θορύβου και είχε προσπαθήσει να μειώσει την ηχορύπανση από τα οχήματα δημοσίας χρήσεως. Ο θόρυβος όμως ε, που μας πλήττει είναι στα 2-3 δεσιμπέλ και υπάρχουν και άλλες πηγές των οποίων η, δυνατότητα φτάνει στα 10 δεσιμπέλ και εδώ θα πρέπει να επηρεάσουμε και να επέμβουμε στην υποδομή. Δηλαδή στις περιφέρειες και τις κοινότητες πρέπει να απευθυνθούμε και γνωρίζουμε ότι η δημοσιονομική θέση των ε, Δήμων και Κοινοτήτων είναι πολύ στενάχωρη και ουσιαστικά ε, πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει στην Ευρώπη. Γι' αυτό και αναρωτιέμαι αν επαρκεί να ζητήσουμε απλώς μία αποδοχή των τύπων οχημάτων ή αν υπάρχουν και άλλοι τομείς τους οποίους θα έπρεπε να εξετάσουμε. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει έρθει ακόμη αλλά θα έρθει και ούτως ή άλλως ε, οι απαντήσεις θα απαντηθούν την άλλη εβδομάδα. Η κυρία Ρούλε, Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια η οποία έχει περιγράψει ε, ποιες είναι οι αρμοδιότητες της, ε, της ε, Επιτροπής μας κατά τρόπον ώστε να μην χρειάζεται να αποδείξουμε στο Συμβούλιο ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Βλέπω ποιο είναι το αρχικό έναυσμα της συζητήσεως για μας που που είναι αξιοπιστία της νομοθεσίας και προστασία των καταναλωτών. Αυτή τη στιγμή ε, δεν μπορώ να ε, σχολιάσω την πρότασή σας την οποία πρέπει πρώτα να διαβάσω και πρέπει να δούμε στη συνέχεια πόσο θα συμπεριφερθούμε και θα συντονιστούμε με την Επιτροπή Περιβάλλοντας και όσον αφορά τον τεχνητό θόρυβο που είναι επίσης αντικείμενο της δικιάς μας Επιτροπής. Ε, με ενδιαφέρει ο θόρυβος των ηλεκτρικών οχημάτων και η μείωση του θορύβου αυτό πρέπει να επιζητηθεί. Δεν πρέπει να αυξήσουμε την ηχορύπα πρέπει να υπάρχει μία λογική ε, εναρμόνιση και να αποφύγουμε τις γελίες εξάρσεις. Ελπίζω λοιπόν ότι θα έχουμε μία καλή συνεργασία. Βλέπω κύριε Μάντερς ότι επανέρχεστε και είναι η κατάλληλη στιγμή. Θέλετε να πάρετε το λόγο αμέσως. Good. Möchten Sie noch ein statement machen? Θέλετε να κάνετε ε, μία, κάποια δήλωση ή εσείς ε, απλώς στηρίζετε ό,τι ελέγχθη, στηρίζετε. Εν τω μεταξύ όμως έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ich glaube, das sollten die später unter sich machen. Ja, Möchte Μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρία Βέστφάλεν θέλετε να επαναλάβετε τα ερωτήματά σας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσει να μας απαντήσει μια και καλή. Ωραία. Ευχαριστώ. Καταρχήν, Δεν θα τα ξαναπώ όλα, αλλά ευχαριστώ για την πρόταση, γιατί όσον αφορά την οδική ε, κυκλοφορία ε, και τον θόρυβο, είναι μία πολύ χρήσιμη πρόταση. Παρόλα αυτά όμως, κατά τη γνώμη μου και για πολλούς ακόμη, τίθενται διάφορα ερωτήματα από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, διότι έχουμε ενημερωθεί και προετοιμαστεί. Καταρχήν αντιλαμβάνομαι ότι η πρόταση βασίζεται στις παλές κατηγορίες αυτοκινήτων και ακούμε από διάφορους τομείς και από την εμπλεκόμενη αυτοκινητοβιομηχανία ότι νέες προτάσεις δεν έχουν συνυπολογιστεί. Μιλάμε για οχήματα του 1985 που είναι ήδη 27 χρονών ε, και ε, ε, ε, και θεωρήθηκαν σαν βάση ενώ τώρα είναι μια ελάχιστη, ένα ελάχιστο ποσοστό των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων και πιστεύουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα αποδώσει νομοθεσία. Θα θέλαμε να ξέρουμε πώς θα προχωρήσει η διαδικασία για τα τεστ, για τις ε, εξετάσεις και δοκιμές, διότι βλέπω ή τουλάχιστον μου ελέγχθη ότι ε, πρέπει κανείς ε, να μεταφέρει τις τάξεις μη ένα, μη δύο, εν δύο, εν τρία ενώ ο θόρυβος αν είστε 125 κιλοβάτα ανατόνο ενώ υπάρχουν άλλα οχήματα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες αυτές μη και νη. Εάν αυτό ισχύει γιατί δεν διατυπώνονται και νέες κατηγορίες οχημάτων. Πιστεύω λοιπόν ότι ένα μεγάλο μέρος η συγχωρυπάνσεως θα μπορούσε να μειωθεί ε, και πιστεύω ότι δεν αναφέρεστε καθόλου στην επίστρωση των δρόμων πράγμα το οποίο αποτελεί μία έλλειψη. Ευχαριστώ και η κυρία Βάις Γκέρμπερ θέλει κάτι να προσθέσει. Δύο ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα ε, τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέει η κυρία Βάις Μπέργκερ. Καταρχήν, όπως η κυρία Βέστφάλεν, πιστεύω ότι ο πίνακας αυτός βασίζεται σε παλιές κατηγορίες αυτοκινήτων και ακριβώς για αυτές τις κατηγορίες και ε, προσέθεσα ε, και ναι, ε, θα ήθελα να ακούσω όμως τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και εμείς θέλουμε να υπάρχει μείωση του θορύβου στην πηγή. Άρα θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και άλλους παράγοντες. Επιπλέον θα ήθελα να ξέρω πώς αξιολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα έπρεπε να υπάρχει μακροπρόθεσμος στόχος με μία μακροπρόθεσμη προοπτική που θα ικανοποιούσε και την αυτοκινητοβιομηχανία και ποια είναι η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σήμανση, η οποία ισχύει για τα ελαστικά, ε, για τις ρόδες. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ε, αν έχει κάποια πρόταση να διατυπώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάποια άλλη νομοθεσία και όσα αναφορά τα ηλεκτρικά οχήματα πρέπει να πούμε ποια, πώς πρέπει να ακούγονται οι θόρυβοι και όχι πώς δεν πρέπει να είναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλοι συνάδελφοι που θέλουν ενδεχομένως να τοποθετηθούν επί του θέματος. Όχι. Ωραία. Τότε δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Merci, Madame la Présidente. Euh, Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλύπτει το σύνολο των οχημάτων. Σημείο κίνησης της πρότασης αυτής είναι μία σειρά δοκιμών που έγιναν για να μπορέσουμε να κάνουμε τη σύγκριση ανάμεσα στην παλαιά ε, μέθοδο ε, για να δούμε πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε το θέμα της ηχοστάθμης που παράγει η μηχανή του οχήματος με την ε, νέα κατάσταση που προσπαθεί να ρυθμίσει συνολικά ε, την ηχοστάθμη των οχημάτων για χρόνια πολλά. Την περίοδο 2000-2005 προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη τις πλέον απτές συνθήκες για να μπορούμε να καταλήξουμε σε μετρήσιμα στοιχεία και να δούμε ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην παλαιά και τη νέα πρόταση. Η νέα πρόταση καλύπτει όλα τα οχήματα. Η κατηγοριοποίηση που αναφέρατε, ναι, πράγματι, η κατηγοριοποίηση στην παλαιά πρόταση υπήρχε. Την αναπαράγαμε μόνο ως οδηγό για να έχουμε ένα σημείο αναφοράς και να μπορούμε να κάνουμε χρήσιμες συγκρίσεις σε σχέση με το πώς μετρούσαμε στο παρελθόν και πώς μετρούμε τώρα. Άρα, να μπορούμε να αναγυγνώσουμε πιο εύκολα το ζήτημα και να δούμε ε, πώς μπορούμε να έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία πάντοτε όσοι να αφορά στην παλιά πρόταση. Για πρακτικούς λόγους. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι το 1985 είχαμε πολύ διαφορετικά οχήματα από αυτά που κυκλοφορούν σήμερα στους δρόμους. Τα οχήματα όμως αυτά δεν υπάρχουν πλέον στους δρόμους σίγουρα. Χρειάζεται όμω ένα πίνοκα για να μπορούμε να κάνουμε συγκρίση ανάμεσα στι παλαιέ τιμές που μετρούσαν την ηχοστάθμη ε, του κινητήρα με τις ε, τιμές ε, πλέον σήμερα που μετρούν το θόρυβο που κάνει το όχημα συνολικά. Το ερώτημα είναι μπορούμε να προσαρμόσουμε τις κατηγορίες με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στα οχήματα που σήμερα ε, διαθέτει η αγορά. Πώς μπορούμε να εξετάσουμε το πώς μπορούμε να ορίσουμε καλύτερες κατηγορίες ώστε να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα σήμερα. Ναι, σωστό αυτό. Ο στόχος πάντως είναι να συνεχίσουμε να έχουμε τις τιμές εκείνες που προτείνει η Κομισιόν ώστε να οδηγηθούμε σε βαθμία μείωση της συγχωρήπανσης. Πρώτο και βασικό στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι η πρόταση αυτή πράγματι καλύπτει τα οχήματα. Δηλαδή δεν καλύπτει την ηχορύπανση που μπορεί να είναι αποτέλεσμα, αν θέλετε, της ποιότητας του οδοστρώματος. Γιατί στη νομική μας βάση δεν μπορούμε, ε, μα, δεν μας επιτρέπει η νομική μας βάση να ασχοληθούμε με κάτι τέτοιο. Χρειάζεται βεβαίως μια σφαιρική προσέγγιση, το πιστεύω και εγώ. Και δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα της χορύπανσης εστιάζοντας μόνο στα αυτοκίνητα. Αυτό το έχει υποθεί πολλές φορές και με τους εκπροσώπους ε, των κυβερνήσεων που είναι αρμόδιοι σε θέματα υποδομών, το έχουμε συζητήσει εκτενώς και υπάρχει σε ένα βαθμό μια συμφωνία πλέον μεταξύ των κρατών μελών ότι η πολιτική μείωση τη συγχώρηπανση περνά από τη μία πλευρά με τη μείωση των εκπομπών ε, των ρήπων των οχημάτων, ναι, αλλά ταυτόχρονα και με την βελτίωση των, του οδοστρώματος ε, και άρα χρειαζόμαστε συγκεκριμένη νομική βάση γι' αυτό. Τώρα, οι προτάσεις της ε, εισηγήτρια είναι πολύ ενδιαφέρουσες, ιδιαίτερα ε, σε ό,τι αφορά την επισήμανση. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συγκεκριμένες πρακτικές για την επισήμανση και ιδίως για την επισήμανση σε θέματα χορύπανσης. Αυτό αφορά και τα ε, λάστιχα των οχημάτων. Υπάρχει μία πρόταση που υποθετήθηκε το 2009 και από ό,τι γνωρίζω από το 2012 ένας από τους στόχους μας πλέον είναι να ολοκληρωθούν οι απαιτήσει σε θέματα ηχορύπανσης που ήδη ισχύουν για τα ελαστικά με βάση την πρόταση του 2009 με την καλύτερη πληροφόρηση του καταναλωτή. Είναι κάτι που δεν εμπεριέχει αρχικά η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά επισημαίνω σε όλους αυτούς τους τομείς και ιδίως στον τομέα των ελαστικών έχουμε κάνει προτάσεις που μπορούν να κινηθούν προς μια κατεύθυνση όπως με την εισηγήτρια. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι οι πιο μακροπρόθεσμοι στόχοι σε αυτό το στάδιο δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθεί τελεσίδικα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρώτη η πρωταρχική μας ανησυχία ήταν η εξή. Θελήσαμε να καταθέσουμε μία πρόταση που θα συνέχιζε το δυναμικό, τη δυναμική εξέλιξη που διακόψαμε εμείς στη δεκαετία του 90. Από το 95 και μετά δεν έχει τεθεί ε, τέτοιο ζήτημα. Είναι μακρά η περίοδος, σχεδόν 17 χρόνια έχουν παρέλθει. Λοιπόν, θέλαμε να συνεχίσουμε αυτή τη δυναμική πορεία και να διασυνδέσουμε ε, αυτή τη διαδικασία με τη νέα μέθοδο δοκιμών. Ε, νομίζω ότι συζητήσεις με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο μέλλον θα προκύψουν διάφορα νέα στοιχεία και θα εξετάσουμε με ποιο τρόπο, ε, ποιο είναι ο καλύτερος τρόπος μάλλον για να οργανώσουμε τις εργασίες με τις εκπομπής, των εκπομπών μάλλον των αυτοκινήτων. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρία Βάις θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω για τη, τα σχόλια και ιδίως για την ειλικρίνεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κατηγορίες. Φαντάζομαι ότι η σύγκριση με τις παλιές κατηγορίες δεν είναι αποφασιστική για τις κατηγορίες τώρα και γι' αυτό θα το δούμε το, όταν θα κοιτάξω την έκθεσή μου που έχω καταρτήσει αγγλικά και απλώς θα ήθελα να με ενημερώσετε σχετικά με αυτές τις κατηγορίες. Χαίρομαι ε, και για τη σήμανση και για τις μακροπρόθεσμες τιμές και όπως σας είπα η επόμενη συζήτηση θα γίνει βάσει της εκθέσεώς μου στις 8 Μαΐου και θα υπάρχει επαρκής χρόνος μέχρι τις τροπολογίες ώστε να, αλλάξουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις ε, με ε, ε, τους συναδέλφους και να δούμε ε, πώς θα προχωρήσουμε για να ε, μπορέσουμε να προβούμε σε μία εναρμόνιση χωρίς να δημιουργήσουμε προβλήματα διότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εσωτερική αγορά. Αυτό τονίζω και προσβλέπω σε μια καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ναι, εδώ θα πρέπει να σας πω ότι η προθεσμία, η συζήτηση μάλλον θα γίνει στις 8 Μαΐου για να έχουμε τις μεταφράσεις και μετά τροπολογίες μέχρι τις 15 Μαΐου το μεσημέρι. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζουμε ότι ε, η αλλαγή θα ξεκινήσει από τις κυρίες που βλέπετε εδώ και το καταλάβατε από τις ευχαριστήσεις ευχαριστήσεις τους. Τώρα πολύ σωστά είμαστε στο, στη συζήτηση και στο χρόνο μας και δίνω το λόγο τώρα στην κυρία Λεγκρή. Η σκιώδης η συγγήτρια θα είναι η κυρία Γκέπχαρτ, μετά ο Όλε Σμίτ απουσιάζει, αλλά η κυρία Λεγκρή έχει πρώτη το λόγο. Euh, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ουσιαστικά εγώ νόμιζα ότι θα αντιδρούσα και θα εξέφρασα τις απόψεις μου σε σχέση με την παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά αντιλαμβάνομαι τώρα ότι ε, εγώ είμαι αυτή που θα πρέπει να παρουσιάσω το θέμα. Ε, πρόκειται για την αναθεώρηση του τελωνιακού κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και θέλουμε να εξετάσουμε τις αδρές γραμμές της μεταρρύθμισης ε, με ένα πρώτο στάδιο. Από την έγκρισή του το 1992 και μέχρι την έγκριση ενός κανονισμού το 2008 δεν είχε μεταρρυθμιστεί ο τελωνιακός κώδικας. Πρόκειται για τον κανονισμό 450 το 2008 που άρχισε να ισχύει στα τέλη Απριλίου το 2008 με στόχο να προσαρμόσουμε τα τελωνία στα ηλεκτρονικά συστήματα και στις νέες ηλεκτρονικές ε, συναλλαγές. Μιλώντας λοιπόν για αυτόν τον κανονισμό του 2008, είχε προβλεφθεί ότι οι εκτελεστικές διατάξεις έπρεπε να εφαρμοστούν ταυτόχρονα με τον ε, κανονισμό. Όπως γράψαμε όμως και αναφέραμε στην έκθεση Σαλβίνη που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο το 2011, η προθεσμία για την οριστικοποίηση των εφαρμοστικών διατάξεων δεν ε, μπορεί να γίνει σεβαστή δεν μπορεί λοιπόν να τηρηθεί κυρίως ε, λόγω των ε, μεγάλης κλίμακος ε, αλλαγών που πρέπει να γίνουν στα ηλεκτρονικά τελωνιακά συστήματα. Αυτός είναι ο βασικός λόγος επίσης. Ταυτόχρονα άρχισε να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παρουσίασε πριν από λίγες εβδομάδες μία τροποποιητική πρόταση του κανονισμού του 2008 αναθεώρησε δηλαδή του τελωνιακού κώδικα Πρωτού καν εφαρμοστεί πλήρως ο κανονισμός ε, του 2008. Είναι λίγο ιδιάζουσα η περίπτωση. Ε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει διάφορους στόχους. Πρώτον, η ημερομηνία θέσης εφαρμογή του τελωνιακού κώδικα επαναπροσδιορίζεται και ο στόχος ε, είναι δυσχερής ακριβώς λόγω των περιορισμών του χρονοδιαγράμματος ε, και επίσης υπάρχουν και διάφορα τυπικά νομικά ζητήματα. Ο νέος κανονισμός που εισηγεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης ως στόχο την προσαρμογή του τελωνιακού κώδικα ε, στα νέα δεδομένα που ισχύουν μετά τη θέση ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας. Υπάρχουν κάποιες προσαρμογές που εκπρόσωπες φαίνονται απλές όπως παραδείγματο χάρη τροποποίηση του κώδικα LBL ε, είναι ο κώδικας ε, των ε, τελωνίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλαγή της φρασιολογία της διατύπωσης μέσα στο διατακτικό του κειμένου ώστε να λάβουμε υπόψη τη νέα σημασιολογία της συνθήκης της Λισαβόνα. Επίσης τίθεται ζήτημα κατανομής αρμοδιοτήτων ανάμεσα δηλαδή στις πράξεις κατεξουσιοδότηση και τι υπόλοιπε εφαρμοστικέ διατάξει άρθρο 290 και 291, τέλος... Άλλος στόχο για της μεταρρύθμισης που μα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το να λάβουμε υπόψη τι εξελίξεις που σχετίζονται με την ασφάλεια, την ε, πρότυποποίηση των ε, ε, συστημάτων, των λειτουργικών συστημάτων πληροφορικών ε, συστημάτων ε, των τελωνίων. Ε, αυτές είναι οι προτινόμενες αλλαγές. Πέραν αυτού, Πέρα από όλε αυτέ τι αλλαγέ και τι ε, προσαρμογέ ε, που απορρέουν ε, από τη θέση σε ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα, υπάρχουν και πολύ πιο ουσιαστικέ προσαρμογέ που τίθενται επιτάπητο τώρα και παρουσιάζονται στο κείμενο 250 σελίδων που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Εντάχει θα διατρέξω κάποιε από αυτέ τι αλλαγέ που θεωρώ εγώ ουσιαστικέ. Δεν έχουμε τον κεντρικό εκτελονισμό μετά από έγκριση των τελωνιακών αρχών επιτρέπεται ε, η τελωνιακή διασάφηση και η καταβολή της τελωνιακής ε, οφειλής στον τελωνιακό σταθμό όπου ε, έχει την έδρα του Οικονομικός Φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανεξαρτήτως που, που, που βρίσκεται ο τελωνιακός σταθμός όπου βρίσκονται τα εμπορεύματα. Μεγάλη πρόοδος, διότι έτσι προωθούμε την ε, σύγκληση των τελωνιακών ε, διαδικασιών ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την κεντρική τον κεντρικό εκτελονισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει βαρκείς πληροφορίες σε σχέση με την ε, εφαρμογή των εφαρμοστικών διατάξεων. Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία. Επίσης, προσωρινή αποθεματοποίηση. Ε, αυτό είναι απαραίτητο για μια καλύτερη εναρμόνιση των τελωνίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις εκτελεστικές διατάξεις σε αυτό το τομέα. Τονίζω επίσης τη σημασία του άρθρου 6 της πρόταση κανονισμού που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άρθρο 6 λοιπόν, απαραίτητο άρθρο για τον εξυγχρονισμό των τελωνίων και προβλέπεται η εξή αρχή. Ε, το ηλεκτρο τα ηλεκτρονικά έγγραφα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως βάση για οποιαδήποτε συναλλαγή ανάμεσα στους εμπορευομένους και τα τελωνία ή τις εθνικές αρχές. Αυτό είναι προφανές διότι χρειαζόμαστε αυτήν την τεκμηρίωση ούτως ώστε να είναι ασφαλείς οι συναλλαγές εμπορευμάτων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πρόταση όμως κανονισμού που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχω την εντύπωση ότι ανοίγεται ο δρόμος για κάποιες εξαιρέσεις που μπορεί να εκφυλίσουν πρωτη ομως κανονισμου που κατεθεσε η ευρωπαικη επιτροπη εχω την βασική αρχή ε, της πρότασης, οπότε θα φροντίσουμε να είμαστε σε γρήγορση ούτω ώστε οι εξαιρέσει να ε, επιτρέπονται σε έκτακτε περιπτώσει ε, και πραγματικά τα, το ηλεκτρονικό υλικό, τα ηλεκτρονικά έγγραφα να είναι η βάση όλων των συναλλαγών ανάμεσα στου εμπορευμένου και τα τελωνία. Επανέρχομαι στα άρθρα 290 και 291 μετά την ε, θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτά τα άρθρα οδηγούν σε έντονες συζητήσεις και σίγουρα η σημερινή μας ε, συζήτηση θα χαρακτηριστεί από τις αψημαχίες που προκύπτουν ε, από αυτήν την αντιπαράθεση ανάμεσα στις πράξεις κατεξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις Ε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε σαφέστατοι για την κατανομή αρμοδιοτήτων άμεσα στι πράξει κατεξουσιοδότηση και τι εκτελεστικέ πράξει, ώστε να μην προκύψει η συμφόρηση κατά την νομοθετική ε, την ε, διαδικασία εκτέλεση των νομοθετικών διατάξεων, είτε σε κάποιο θεσμικό όργανο, είτε γενικότερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το χρονοδιάγραμμα τώρα. Μέσα στην πρόταση τροπή του κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν προβλέπει ότι ε, πριν από τις 24 Ιουνίου 2013 οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουν τεθεί σε ισχύ ε, αυτές οι διατάξεις ε, και στους 18 μήνες μετά τη θέση σε ισχύ του κανονισμού, μετά τον Ιούνιο το 2013, δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο 2014 πρέπει να έχουν τεθεί σε ισχύ οι εφαρμοστικές διατάξεις με στόχο την ευθυγράμμιση των συστημάτων πληροφορικής. Βάσει του προγράμματος της Επιτροπής, η προθεσμία για την θέση σε λειτουργία αυτών καθεαυτών των συστημάτων πληροφορικής έχει τεθεί την 31η Δεκεμβρίου του 2020. Το ίδιο ισχύει και για την επιγραμμική λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων. Βεβαίως... Ε, εάν καθυστερήσουμε και λόγω της διαρκούς τεχνολογικής εξέλιξης αυτών των συστημάτων πληροφορικής ε, θα καταπέσει η ίδια η πρόταση γιατί δεν θα είναι πλέον εφαρμόσιμη. Είναι εξαιρετικά τεχνικό ε, και περίπλοκο το ζήτημα και σχετίζεται με την ίδια τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Άρα όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να διακατέχονται από ένα θετικό και επικοδομητικό πνεύμα, ούτω ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε το ίδιο από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου, δηλαδή να είναι ενεργό η εταιρική αυτή σχέση που έχουμε. Ταυτόχρονα μην ξεχνάτε ότι επεξεργαζόμαστε και ε, το οικονομικό το ε, κομμάτι ε, των τελωνίων, το πρόγραμμα Φίσκους και αυτό περιπλέκει ακόμη περισσότερο τις ε, εργασίες μας. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση λοιπόν για την τήρηση των ε, προθεσμιών που έχουν τεθεί στο χρονοδιάγραμμα να μην χαθούμε σε μικρές ε, διαθεσμικές διενέξεις και χάσουμε το χρόνο γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα και θα πρέπει να αυτοπιθαρχηθούμε. Ευχαριστώ την κυρία Λεγκρίπ. Η κυρία Γκέπχαρ τώρα έχει το λόγο. Ε, θέλω να ζητήσω συγγνώμη την ε, συνάδελφο Σιλβάνα Ράπτη που έχει ραντεβού στην Ελλάδα και χρειάστηκε να φύγει απρόοπτος. Μου έχει αφήσει όμως τα ε, σχόλιά της τα οποία ευχαρίστως θα παρουσιάσω είναι, ε, είναι γραμμένα μεν αγγλικά αλλά θα προσπαθήσω γιατί έχω πολύ κακή προφορά αγγλικά να τα διαβάσω γερμανικά αποβλέπει εις ε, την βελτίωση του τελωνιακού κώδικα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, και στην ε, έκθεση του περασμένου Δεκεμβρίου η Επιτροπή είχε αντιληφθεί ότι έχει πρόβλημα για μία σύντομη υλοποίηση της αναμορφώσεως του τελωνιακού κώδικα και δεν θα μπορέσει να γίνει σεβαστή η ημερομηνία του 2013 διότι ε, χρειάζονται τεχνικές προσαρμογές ε, πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση των εμπλεκομένων και ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα και όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα και δεν μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα. Αντιλαμβάνεται λοιπόν αυτές ε, τις δυσκολίες αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να σηκώσουμε τα χέρια και ξέραμε από την αρχή ότι μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες οι οποίες είχαν συνυπολογιστεί. Γι' αυτό και καλεί η κυρία Ράπτη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να μας πει γιατί από τόμος υπάρχουν νέα στοιχεία για την εφαρμογή του τελωνιακού κώδικα διότι αν κατάλαβε καλά ε, τώρα προτείνεται το έτος ε, εφαρμογής 2020. Αν ευσταθεί αυτό για ποιο λόγο και για, ποιους, ε, για ποιες αιτίες έχει προταθεί αυτή η ημερομηνία. Εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε να υπάρχουν υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας και μία σύντομη και σύμφωνα με τις διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε διατηρήσει σαν έτος πιθανής εφαρμογής του νέου τελωνιακού κώδικα το 2016, δηλαδή 7 χρόνια αργότερα από αυτό το οποίο υπήρχε στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 4 χρόνια το, μάλλον είναι 7 χρόνια αργότερα από την αρχική επιτροπή της, από την αρχική πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2020 αναφέρουμε και 4 χρόνια αργότερα από αυτό που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί λοιπόν αμφισβητείτε αυτή η πρόοδος, πώς σκοπεύετε να μας απαντήσετε, διότι υπάρχουν υπάρχουν και διάφορα θέματα τα οποία πρέπει να αξιολογήσουμε θετικά, δηλαδή αντί για την επιτροπολογία εξουσιοδότηση πράξης, ε, μία προσαρμογή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή στην εργασία αυτή, και ε, όλα αυτά τα θέματα είχαν θυγεί ε, ήδη στην πρώτη εφαρμογή του τελωνιακού κώδικα και τότε πρέπει να αξιολογηθούν για να δούμε ε, πώς επηρεάζουν και γι' αυτό να καταρτιστούν οι αναγκαίες τροπολογίες. Ευχαριστή την κυρία Λεγκρή για την καλή συνεργασία στον τομέα αυτό και με αυτά εγώ κλείνω τα σχόλια που έκανα εν ονόματι της συναδέλφου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Όλε Σμιτ των Φιλελευθέρων τώρα. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη που αργοπόρησα. Είστε, είστε όλοι πολύ γρήγοροι εδώ. Καλό είναι αυτό. Το βασικό για μένα και το είπε και η κυρία Γκέφχαρτ είναι το χρονοδιάγραμμα. Το είπε και η συγγήτριά μας. Νομίζω ότι είναι δύσκολο για κάποιους να καταλάβουν γιατί πρέπει να περιμένουμε τόσο πολύ καιρό. Εφόσον εκπροσωπείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έπρεπε ο εκπρόσωπος να μας εξηγήσει γιατί ε, προβλέπεται ε, τέτοια μεγάλη ε, καθυστέρηση, κάτι που συμβαίνει και σε σχέση με άλλα νομοθετήματα. Νομίζω, ζητώ συγγνώμη που ξεκινάω με κάτι δυσάρεστο, αλλά ή, αν δεν τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα δεν θα μπορέσουμε καν να προχωρήσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το σχέδιο. Τώρα κάτι άλλο. Καταλαβαίνω ότι δεν, έχουν, δεν δέχονται όλα τα κράτη-μέλη ε, ε, να υιοθετήσουν το νέο σύστημα και η εισηγήτρια νομίζω αναφέρθηκε σε αυτό. Δεν χρησιμοποιούν τις κοινέ ε, πλατφόρμες και τα υπόλοιπα εργαλεία πληροφορικής που τους προτείνονται. Κάποιες χώρες δεν το δέχονται και θα μπορούσατε ίσως να με ενημερώσετε για αυτό το θέμα. Έχετε περισσότερες πληροφορίες. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε επίσης για να καλύψουμε αυτό το κενό, να αναπληρώσουμε το χρόνο που μας λείπει. Τι, ποιο είναι το πρόβλημα, ο προϋπολογισμός είναι, πώς μπορούμε να επισπεύσουμε τη διαδικασία. Και τρίτον, Ε, και αυτό είναι πάντοτε ένα ε, λεπτό ε, πολιτικό ζήτημα πρόκειται για την ηλεκτρονική αποθήκευση των πληροφοριών. Άρθρο 7. Πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Θα έχει την ερμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει πράξεις κατά εξουσιοδότηση που θα προσδιορίζουν τους κανόνες σχετικά με την αποθήκευση των δεδομένων. την περασμένη εβδομάδα ψηφίσαμε για τα στοιχεία επιβατών, τα PNR. Το ξέρετε και ξέρετε και πόσο λεπτό ήταν το ζήτημα. Τι πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως ε, το Συμβούλιο πώς ε, τοποθετείται σε σχέση με αυτό το τόσο ε, ευαίσθητο από πολιτική σκοπιά ζήτημα. Κατά τα λοιπά, προσβλέπω στη συνεργασία με την εισηγήτρια. Πιστεύω θα είναι χρήσιμο, αλλά επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ κρίμα που πρέπει να περιμένουμε τόσα χρόνια για να εφαρμόσει το σύστημα. Ευχαριστώ τον Όλε Σμιτ. Εν τω μεταξύ ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορώ να σας πω ήδη ότι όλοι ήθελαν να ρωτήσουν γιατί το χρονοδιάγραμμα έχει διαρκέσει τόσο χρόνο και τώρα παίρνω τους επόμενους σκιώδεις για τους πρασίνους υποθέτω η κυρία Ρούλε. Ε, ευχαριστώ. Συμφωνώ με τα σχόλια του Όλε Σμιτ διότι και εγώ ανησυχώ σιγά σιγά σχετικά με αυτή την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος όσο αναφορά τα στοιχεία και την ανταλλαγή στοιχείων θέλω να ρωτήσω αν ε, έχει ληφθεί υπόψη και η γνώμη του υπευθύνου προστασίας των δεδομένων διότι έχουμε πρόβλημα με το θέμα αυτό και θα ήθελα να ε, ζητήσω από τον υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων γιατί υπάρχει αυτό το έλλειμμα θέλημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Άλλοι σκιώδεις παρίστανται από το ECR, άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι θέλουν να παρέμβουν. Διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ξεκινήσει με την απάντηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ζητήσω συγγνώμη, διότι μόλις έφτασα, αλλά δεν με είχαν ενημερώσει ότι προχωρούσα τόσο γρήγορα και άκουσα μόνο ε, τα, την τελευταία παρέμβαση του κυρίου Σμιτ για ε, τη κυρία ε, Ρούλε, δηλαδή των δύο σκιωδών από τις τελευταίες πολιτικές ομάδε που τοποθετήθηκαν. Δυστυχώ δεν άκουσα όλα τα υπόλοιπα σχόλια, όλη την υπόλοιπη συζήτηση. Ζήτω συγγνώμη. Δεν μπόρεσα να κάνω την παρουσίασή μου στην ε, έναρξη της συζήτησης. Δεν ξέρω, ε, Πρόεδρε, θέλετε να κάνω την παρουσίαση παρόλα αυτά, γιατί έχω την εντύπωση ότι ε, θα μας διαφωτίσει η παρουσίαση για διάφορα σημεία που σχολίασαν οι εισηγητές ως προς την ηλεκτρονική διάσταση της εφαρμογής του τροποποιημένου κανονισμού των τελωνίων. Θα, τα μιλήσω, θα μιλήσω στα αγγλικά γιατί ήταν η παρουσίασή μου στα αγγλικά, την έχω συντάξει στα αγγλικά. Βασιζόμαστε σε έναν ε, υφιστάμενο κανονισμό, το 450 του 2008, ε, που προβλέπει τα περί εξυγχρονισμένου τελωνιακού κώδικα. Η πρόταση που τώρα εξετάζουμε προβλέπει αναθεώρηση του κανονισμού 450 και ξέρουμε ότι οι τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους προτείνεται αναθεώρηση είναι ε, οι εξή ε, και αναφέρουμε σε αυτά που είπαν οι σκιώδεις εισηγητές. Πρώτον, πρέπει να ε, δούμε αν τον Ιούνιο του 2013 θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός το 2008 και να καταλάβουμε ποιες θα ήταν οι συνέπειες. Δηλαδή, για το εμπόριο και για τη τελωνία, ε, ο στόχο ήταν να μην έχουμε καθόλου χαρτί, ε, καθόλου έγγραφα, αλλά συνειδητοποιήσαμε ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει το σύστημα και προσπαθήσαμε με διαβούλευση όλων των φορέων, οικονομική φορή, τελωνία κτλ. Συζητήσαμε ε, όλε τι πιθανέ λύσει πληροφορικής και τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής. Δεύτερος λόγος ε, τήρηση της δέσμευσης που έχει να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περί ευθυγράμμισης αυτού του κανονισμού που ήδη ήταν ευθυγραμμισμένος με τη διαδικασία εξέτασης ε, με την συνθήκη της Λισαβόνας για το δύο θέματα, δηλαδή της πράξης κατεξοσοδότησης και τις εκτελεστικές πράξεις. Ε, τρίτο, αλλά σημαντικό, από το 2008 και μετά Ω προ τον εξυγχρονισμό του τελωνιακού κώδικα και την περιγραφή των ε, διαδικασιών που θα πρέπει να θεσπιστούν, κρίναμε όλοι μαζί και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί ότι χρειάζονται προσαρμογέ για κάποιε διατάξει, ούτω ώστε να λειτουργούν και μάλιστα με αποτελεσματικό τρόπο στην πράξη. Έγιναν ε, ανταλλαγές ε, ανάμεσα στον Επίτροπο Σεμέτα και τον Πρόεδρο της Επιτροπής σας παρουσία φυσικά του, της Προεδρίας του Συμβουλίου για να καταλάβουμε ε, πώς μπορούμε να δράσουμε ταχύτατα. Είναι επίγον. Έχουμε μία ημερομηνία που πρέπει να σεβαστούμε, Ιούνιος 2013. Και να μην ξεχνάμε ότι ο απότερος στόχος είναι να μην ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας, δηλαδή να καταπολεμήσουμε τον πειρασμό, να αγγίξουμε ε, τμήματα του ε, ε, τελωνιακού κώδικα που οι υποφυσιολογικέ συνθήκες δεν θα τροποποιούνταν. Ο στόχος κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτό το νέο, αυτή η νέα νομοθετική πρόταση όταν εφαρμοστεί να λειτουργήσει υπό τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες και με αποτελεσματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικροτεί το ότι υποστηρίχθηκε ο στόχος αυτός ε, μέσα στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 1ης Ενάτου του 2011 με αντικείμενο φυσικά τον εξχρονισμό του τελωνιακού κώδικα. Σε σχέση με την πρώτη προτινόμενη αλλαγή είναι απαραίτητο να αναβάλουμε την θέση εφαρμογή του τελωνιακού κώδικα. Αυτό αναγνωρίστηκε επίσης ε, ω αληθέ από τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Όχι εσάι να, το, να αναβάλουμε την εφαρμογή, αλλά όσο χρειάζεται ώστε να επιτύχουμε ε, με καλύτερο εντοπισμό και κάλυψη των αναγκών μέσω από μέσα από νέα συστήματα πληροφορικής. Από τη, θέση, από την ημερομηνία θέση εφαρμογή του αναθεωρημένου κανονισμού και μετά, οι 18 μήνες μετά συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει εφαρμοστεί και η υπόλοιπη διαδικασία, δηλαδή να έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τότε όλες τις πράξεις κατεξουσιοδότηση. Η θέση εφαρμογή προβλέπεται 18 μήνες μετά τη θέση σε ισχύ. Ε, το πρόβλημα είναι τα συστήματα πληροφορικής, γιατί ένα κράτος μέλος και αρμόδιες αρχές δεν μπορούν να αναπτύξουν σε καμία περίπτωση τα νέα συστήματα πληροφορικής με μιας. Για να οργανώσουμε την ανάπτυξη των νέων συστημάτων ναι, πληροφορικής ε, ε, φτιάξαμε ένα master plan ε, για τα συστήματα πληροφορικής, ένα στρατηγικό σχέδιο και θα λάβετε και τη σύντομη εκδοχή για να δείτε τι θα γίνει, όχι μόνο σε επίπεδο Ένωσης και Επιτροπής, αλλά τι θα γίνει γενικώ ακόμη και στο επίπεδο των χρηστών, το... με τα κράτη-μέλη. Αυτό το master plan θα επισυναυθεί στο πολιετές στρατηγικό σχέδιο το επωνομαζόμενο που θα εγκριθεί και θα δημοσιευθεί για, ε, με υποστηρικτικό ε, ρόλο για την εφαρμογή ε, δηλαδή των αποφάσεων για τα ηλεκτρονικά τελωνία. Στο άρθρο 17 εδάφιο 1 βλέπετε εκεί ότι μεταξύ άλλων προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το συγκεκριμένο στόχο εξυγχρόνησης του τελωνιακού κώδικα υιοθετείται ένα πρόγραμμα εργασίας ε, που με συμμετοχή των κρατών μελών βάσει της διαδικασία επιτροπολογίας ούτω ώστε να προετοιμαστεί η εφαρμογή υιοθετώντα ε, ε, τις προσφορότερες νομικές διατάξεις και τις καταλληλότερες προθεσμίες εφαρμογής καθώς και τις μεταβατικές περιόδους. Χρειαζόμαστε μεταβατικές περιόδους ούτω ώστε σταδιακά να εφαρμοστούν όλες οι διαδικασίες μέχρι το Δεκέμβριο του 2020 Και αυτό ε, θα συμπέσει με την ανάπτυξη των νέων προγραμμάτων ε, για το φίσκους. Ε, δεύτερο θέμα, η ευθυγράμμιση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά είχε αναλάβει δέσμευση να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της συνθήκης της Λιλεφώνης για την Επιτροπολογία και τις πράξεις κατεξουσιοδότηση. Είχε την πρόθεση να βασιστεί φυσικά στον υφιστάμενο κανονισμό ούτως ώστε να προσδιορίσει επακριβώ το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο των πράξεων κατά εξουσιοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των νέων της αρμοδιοτήτων. οι ανάγκες της εφαρμογής θα καλυφθούν ε, ενδεχομένως και από νέες ε, προσαρμογές της διατάξης. Ε, Χρειάζονται λοιπόν αλλαγές ε, όπως αναφέρει και ο κύριος Σαλβίνη στην έκθεσή του στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον εξυγχρονισμένο τελωνιακό κώδικα. Υπάρχουν και άλλες βελτιώσεις που επιδέχεται η πρόταση, παραδείγματος χάρη διατάξεις για κεντρικό εκτελενισμό για προσωρινή αποθεματοποίηση για τη χρήση κριτηρίων ε, για τους ε, εξουσιοδοτημένους οικονομικούς φορείς που θα μπορούν να ζητούν ειδική έγκριση. Αυτές είναι κάποιες ε, από τις στοιχείες που θα πρέπει να προσαρμόσουμε. Λοιπόν, ε, ε, πρόκειται για μια ειδική διαδικασία αυτή της ε, τροποποίησης του σχεδίου κανονισμού. Χρησιμοποιούμε ένα μοντέλο συνήθως και φυσικά το τηρήσαμε και αυτή τη φορά, αλλά... Ε, σε κάθε περίπτωση έχουμε σωματώσει τις ε, επιθυμητές προσαρμογές. Για να κλείσω θα έλεγα... Αυτή η παρουσίαση έχει σκοπό να βοηθήσει και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για να λειτουργήσει ως ε, εργαλείο. Υπάρχει βεβαίω και πίνακα αντιστοίχηση στην πρόταση. Και υπάρχει και όλη κατάλληλη τεκμήριωση ώστε να μπορούν να εντοπιστούν καλύτερα ποιε είναι οι αλλαγέ που προτείνουμε και, για, και εξηγούμε σε ένα non-paper τι διαδικασία ακολουθήσαμε για να ευθυγραμμιστούμε με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και πέραν αυτού και παράλληλα με αυτό, είπα και πριν, η δουλειά επί του master plan και η δουλειά σε επίπεδο πληροφορικής θα πρέπει να συνεχιστεί παράλληλα. Εν κατακλείδη, οι βασικές αλλαγές που προτείνει η Κομισιόν στην αδιατύπωση του κανονισμού είναι οι νέες ημερομηνίε εφαρμογής του κανονισμού μαζί με τη δέσμευση για την εκπόνηση ενός προγράμματος πληροφορικής, προγράμματος IT, που θα προβλέπει συγκεκριμένο σχεδιασμό και θα ε, προβλέπει και τις κατάλληλες νομικές διατάξεις. Επίσης, σε ευθυγράμμιση με τη συνθήκη βεβαίως, αν δείτε τον αριθμό των αλλαγών, αυτό είναι το αποτέλεσμα της ανάγκης ευθυγράμμισης βάσει των άρθρων 290 και 291 της συνθήκης. Και τέλος, σε ό,τι αφορά τις προσαρμογές, προσπαθήσαμε να τις συνδέσουμε με τα απολύτως αναγκαία για να επιτύχουμε τους ε, στόχους και τις βασικές διαστάσεις ε, και στόχους ε, της, ε, του κανονισμού του 2008. Ευχαριστώ πολύ. Ja, Ευχαριστώ. Νομίζω ότι υπήρξαν ορισμένες διευκρινήσεις. Επανέρχομαι όμως πάλι στο θέμα του αν ε, ε, απαντήσατε στο θέμα του επιτετραμένου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δεν ξέρω αν έχετε ρωτήσει σχετικά με την παρουσία Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μήπως τότε μπορούμε, μπορείτε να επέμβετε να μας διευκρινίσετε το σημείο αυτό για τον υπεύθυνο για τα προσωπικά δεδομένα που ετέθηκε ερώτηση. Ναι, νομίζω όταν μιλάμε για αρχή ελέγχου, ουσιαστικά είναι η αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων. Στο βαθμό που η πρότασή μας είναι μια πρόταση αναδιατύπωση του κανονισμού, η προστασία δεδομένων στα συστήματα πληροφορικής είναι κάτι που δεν αλλάζει τίποτα στην αρχική πρόταση. Προβλέπει μόνο και μια επίσημη διαβούλευση. Στην υλοποίηση τώρα αυτού του νέου κανονισμού, σαν διατύπωση ουσιαστικά, θα πρέπει να υπάρχουν ειδικά συστήματα, ειδικέ καθορισμένες βάσει δεδομένων και θα ορίζεται το σύστημα αυτό με βάση αυτό που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να υπάρχει πρώτα απ' όλα η σχετική γνωμοδότηση του EDPS, της Ευρωπαϊκής Αρχής Προστασίας Δεδομένων. Ähm, Ευχαριστώ. Η κυρία Λεγκρίπ δεν ζητάει τώρα να παρέμβει, οπότε η επόμενη ημερομηνία είναι ε, συζήτηση και πάλι στην Επιτροπή στις 30 Μαΐου και στη συνέχεια 20 Αυγούστου, 17 Οκτωβρίου θα ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό εδώ. Ευχαριστώ για το θέμα αυτό και το τελευταίο εφόσον είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή όλοι έχουμε είμαστε λίγο μπροστά στην ημερήσια διάταξη. Ερχόμαστε τώρα σε ένα σημαντικό θέμα της εργασίας μας, την 20η πέτειο της Ευρωπαϊκής Ενίας Αγοράς και θα μας παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μία παρουσίαση. Bitte? Yes, darum, darum habe ich es äh, gemerkt. Es ist, äh, wir werden uns noch daran gewöhnen müssen, mit dem neuen. Πρέπει να συνηθίσουμε να προσαρμοζόμαστε στο νέο πρόγραμμα και οι συντονιστές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι την ε, πέμπτη το απόγευμα δεν θέλουμε να έχουμε εδώ σε άδεια έδρανα μία συζήτηση και ε, στο τέλος του χρόνου μετά έχουμε πέμπτη απόγευμα πολλές φορές συνεδριάσεις αλλά όσοι θα είναι εδώ θα το αντέξουν τι να κάνουμε και δίνω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την Επιτροπή ΙΜΚΟ που μας δίνει αυτή την ευκαιρία να παρουσιάσουμε εντάχει ένα από τα project τα οποία προωθούμε στα πλαίσια της 20ης επαιτίου της ενιαίας αγοράς γενιά 1992. Ειδικά το φθινόπορο Αναπτύξαμε μια σειρά δράσεων στους κόλπους Επιτροπής και με τη βοήθεια του Κοινοβουλίου για να εορτάσουμε την επέτειο των 20 ετών της δημιουργίας ενιαίας αγοράς. Ο σκοπός δεν είναι τόσο πολύ να γιορτάσουμε την ε, ενιαία αγορά ως αυτή, αλλά για να θυμηθούμε αυτή τη στιγμή ε, και γιατί η ενιαία αγορά είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για να δοθεί μια νέα πνοή σήμερα στην ε, ευρωπαϊκή αγορά ε, και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Δηλαδή δεν θέλουμε απλά ως νοσταλγή να αναπολούμε το παρελθόν, αλλά να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε μια δυναμική στην ευρωπαϊκή οικονομία αυτή τη στιγμή της κρίσης. Τώρα, η γενιά του 1992 επίσης είναι κάτι σημαντικό, γιατί ε, είναι η ενεργοί άνθρωποι σήμερα που ήταν νεότατοι την εποχή εκείνη. Λοιπόν, ο γενικός στόχος της εκστρατείας μας ε, για να γιορτάσουμε αυτήν την επέτειο είναι να θυμηθούν πρώτα απ' όλα τα επιτεύγματα. του στόχου ε, για την ανάπτυξη ε, και να θυμηθούν αυτοί οι νέοι ενήλικε του 1992 ποιοι ήταν οι στόχοι και οι φιλοδοξίες τότε. Αυτή η γενική διαφάνεια σας δίνει μια γενική εικόνα των διάφορων δράσεων που θα αναλάβουμε. Κάτω αριστερά βλέπετε ε, δημοσιεύσεις σε χαρτί και online. Πρώτον, για να θυμηθούμε τα επιτεύγματα, είναι σημαντικό να θυμόμαστε το πριν και το μετά πιο πολλά ευρωπαϊκά δικαιώματα εν προκειμένου, κάτι που μας ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είχε ζητήσει έναν πρακτικό οδηγό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Έπειτα στις 15 Οκτωβρίου θα γιορτάσουμε την εβδομάδα της ενίας αγοράς αλλά και θα γιορτάσουμε και ειδικά την 15η Οκτωβρίου εδώ στις Βρυξέλλες και χαιρόμεθα ιδιαίτερα και το Κοινοβούλιο προσέφερε ε, την αίθουσα της Ολομελίας για να κάνουμε αυτή τη γιορτή. Επίση, το Νοέμβρη θα έχουμε ε, ένα βίντεο το οποίο ελπίζουμε να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά με τη βοήθειά σας και με τις υπηρεσίες σας, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την περίοδο Ιούλιο ως Οκτώβριο θα κάνουμε κάποια κοινά σεμινάρια με αντικείμενο την ε, νέα αγορά. Και εκεί περιμένουμε δραστήρια συμμετοχή των μελών σας. Έπειτα, μέτρα που θα υιοθετηθούν πριν την εβδομάδα της νέας αγοράς και θα γραφήσουν την όλη συζήτηση που θα λάβει η χώρα εκείνη την εβδομάδα. Σε αυτή την διαφάνεια θα δείτε το χρονοδιάγραμμα. Δεν θα το διατρέξω τώρα, δείτε το. Σας παραπέμπω πάλι στο project Γενιά 1992 που ήδη έχουμε λανσάρει, οπότε για να δούμε την επόμενη διαφάνεια. Η Γενιά 1992 τη λανσάραμε πριν από δύο εβδομάδες. Είμαστε λοιπόν στα πρώτα στάδια αυτού του project, το οποίο θα τρέξει έως το Σεπτέμβρη. Οι νικητέ αυτού του project, γιατί είναι ένας διαγωνισμός ουσιαστικά, είναι να συλλέξουμε απόψεις και εμπειρίες των νέων ενηλίκων από την νέα αγορά. Οι νικητέ λοιπόν θα συμμετάσχουν στι εθνικέ εκδηλώσει ε, για τον εορτασμό τη αγορά και φυσικά θα συμμετέχουν και εδώ στην εβδομάδα που, της 15 Οκτωβρίου τη Βρυξέλλες. Έπειτα μετά, να πω ότι ξεκινήσαμε ένα διαγωνισμό για 20χρονους, δηλαδή μόνο όσοι γεννήθηκαν το 1992 μπορούν να συμμετάσχουν. Βεβαίως αποκλείονται πάρα πολλοί και σημαντικοί που θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν και γεννήθηκαν το 1991 και το 1993. Αλλά συναισθηματικά και συγκινησιακά είναι σημαντικό να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό άνθρωποι που γεννήθηκαν το 1992. Οι πιο πολλοί, που το σκεφτήκαμε, είχαμε γεννηθεί πολύ νωρίτερα. Αλλά τι να κάνουμε η ομάδα στόχο δεν είναι μόνο σπουδαστέ, αν και λογικά είναι σπουδαστέ, αλλά προσπαθήσαμε να βρούμε και επιχειρηματίε. Να δείξουμε ποιοι είναι αυτοί οι νέοι 20 έχουν επιχειρηματίε στην Ευρώπη, άνθρωποι που μόλις ξεκινήσαν την καριέρα τους, αλλά και νέου ανέργου που θέλουν να συμμετάσχουν ενεργά στην ε, κοινότητα αυτή, στην ενιαία αγορά. Στόχο, Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Συλλογή απόψεων. Με διάφορους τρόπους εγρήγορση μεταξύ των νέων και εγρήγορση ειδικά για τις ευκαιρίες, όπως επίσης και την ενεργό συμμετοχή του στην διαδικασία α, εντοπισμού των ελλημάτων. Προσπαθούμε και εμείς να εντοπίσουμε τα πρακτικά εμπόδια ε, και τα ελλείμματα μπορούν να καλυφθούν με νέε πολιτικέ στην αγορά. Τώρα, μετά τον Οκτώβριο, μετά από αυτό το project, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτή την πλατφόρμα για περαιτέρω συζήτηση ε, με την ευκαιρία που δημιουργεί για αυτού του νέου ενήλικε. Στην επόμενη διαφάνεια, βλέπετε ότι ο διαγωνισμό είναι ένα δημιουργικό διαγωνισμό με πολλέ μορφέ. Ε, μπορούν να συμμετάσχουν οι νέοι με ένα άρθρο που μπορούν να γράψουν με τι εμπειρίε, απόψει ή να φτιάξουν ένα βιντεάκι για το ίντερνετ ή να κάνουν μια γελιογραφία, ένα καρτούν κτλ. Δημιουργικός λοιπόν διαγωνισμός. Η δημιουργικότητα λοιπόν είναι, αν θέλετε, ε, ο γνώμονας επιλογής των νικητών, αλλά μέσω δημιουργικότητας να μπούμε στην ουσία και να εστιάσουμε στην ουσία τη ενιαίας αγοράς και να προσπαθήσουμε να εκμεύσουμε απόψεις για το πώς βλέπουν οι νέοι ενήλικες την ενιαία αγορά και θα του καλέσουμε λοιπόν να εστιάσουν σε μια σειρά από θεματικές ενότητες, εκπαίδευση, α, συμμετοχή στα κοινά, επιχειρηματικότητα, θέσει εργασία, θέματα πολιτισμού και ψυχαγωγία, ε, πνευματική ιδιοκτησία, περιβάλλον και καταναλωτέ ψηφιακή ενιαγορά, ηλεκτρονικό εμπόριο και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει κανείς στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ε, θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε αυτό το διαγωνισμό με πολλούς τρόπους, με τα κοινωνικά μέσα, στο διαδίκτυο ιδίω, αλλά θα κινητοποιήσουμε και διάφορους μέντορες, οι μέντορες που έχουν εμπειρία. Είναι δηλαδή άνθρωποι στα 28, 30, 32 και σε αυτήν την ηλικία με επιχειρηματική και εργασιακή εμπειρία. Επίσης είναι οι εταίροι, εταίροι του ιδιωτικού τομέα και εκπρόσωποι κοινωνίας των πολιτών για να διαδώσουν, αν θέλετε, αυτή την πρωτοβουλία. Επίσης υπάρχουν και συνάδελφοι από άλλες γαμαδέλτες, όπως είναι η νεολαία σε κίνηση, το Youth on the Move, που μπορεί να βοηθήσει. Νικητέ, πάμε στα στη διαφάνεια. Θα υπάρξει ένα πάνελ κριτική επιτροπή για να επιλέξουν όχι μόνο με βάση τη δημιουργικότητα αλλά και επί τη ουσία. Και θα συμμετάσχουν βεβαίω, οι νικητέ, στι εκδηλώσει τη εβδομάδα ε, του Οκτωβρίου τη Βρυξέλλε. Εδώ λοιπόν στο ημικύκλιο τη Ολομέλεια είναι καλό να έχουμε αυτού του νέου ανθρώπου να μπορέσουν να ανταλλάξουν απόψει με αυτού που χαράσουν πολιτική και να ανταλλάξουν απόψει για το πώ θα θέλουν να βλέπουν την νέα αγορά την επόμενη 20 ετία βραβεία. Βλέπετε εδώ πέρα τα διάφορα βραβεία και ειδικά οι μαθητείες, έτσι είναι κομμάτι των βραβείων, διότι αυτός ο διαγωνισμός θα θέλαμε να πάρει και μια άλλη χρειά. Δηλαδή, όχι να δούμε ποιος μπορεί να κάνει το πιο έξυπνο βιντεάκι, αλλά ποιος θα μπορούσε να ξεκινήσει μια καριέρα, μια σταδιοδρομία, ε, προσφέροντά του μια μαθητεία. Στο τέλος, τι μπορείτε να κάνετε εσείς ε, ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρώτα απ' όλα να συστήσετε αυτήν την ιστοσελίδα, να μιλήσετε στους α, ε, α, ψηφοφόρους σας, στην εκλογική σας περιφέρεια, να μιλήσετε με ε, οργανώσεις νεολαίας, να διοργανώσετε και εσείς με τη σειρά σας τα τις μαθητείες που θα μπορούσαν να κάνουν νικητές και φυσικά, αν έχετε σχετικές δημοσιεύσεις, ε, μπορείτε και εσείς να μας βοηθήσετε για να ε, διαφημίσουμε την εκδήλωση. Πιστεύω ότι αν όλοι από κοινού, η Κομισιόν, οι Ευρωβουλευτές ε, και τα κράτη-μέλη κάνουν αυτή την κοινή προσπάθεια, θα έχουμε να επιτύχει πολλά, διότι η νέα αγορά είναι το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ για την προσοχή και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Είναι καλό που το ξέρουμε εν και υπάρχει και μια ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει καταρτήσει και άλλες προτάσεις και νομίζω ότι ακόμη και αν το διατυπώσατε διστακτικά νομίζω ότι τα επιτεύγματά μας είναι κάτι που πρέπει να ενημερώσουμε για τα τελευταία 20 χρόνια ιδίω τώρα που υπάρχει μία τάση να σηκώσει πάλι κανείς νέους φραγμούς. Ξεκινά όμως η συζήτηση. Αυτή τη στιγμή το ΕΛΚ έχει κάποιον εκπρόσωπο. Ήθελα να πάμε κατά σειράν ή από πλευράς ομορφιάς ή ό,τι επιθυμείτε. Γενιά 92. Μου άρεσε αυτή η ιδέα του στάζ της ε, πρακτικής άσκησης. Στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΜΑΡΚ το συζητήσαμε, αλλά δεν αναφερθήκαμε στο ΣΤΑΖ. Μ' άρεσε η ιδέα. Και από ό,τι κατάλαβα, χρειαζόμαστε στενή συνεργασία. Εσείς προσφέρετε τέτοιες πρακτικές ασκήσεις. Εμείς πάντως ναι. Α, και εσείς. Ωραία. value, if... Τότε να συνεργαστούμε για να έχουμε προστιθέμενη αξία. Μπορούμε να προσφέρουμε ε, πρακτικές ασκήσεις ε, ε, στους 20χρονους που έτσι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό αυτό και από ό,τι κατάλαβα θέλετε αυτό να είναι και ο πυρήνα τη εκδήλωση που θα γίνει στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή, πολλή ενέργεια, πολλοί νέοι, να δοθεί μια δυναμική στη διαδικασία. Αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας και κινητοποιήσουμε τους συναδέλφους, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Χρειάζεται προώθηση όμως, διαφήμιση. Δεν το βλέπουμε, δεν τη βλέπουμε τη γενιά το 92 πουθενά στο διαδίκτυο σχεδόν. Χρειάζεται μια σοβαρή ε, και μαζική εκστατεία ενημέρωσης. Η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι αναφέρεται ότι έχει γίνει και θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον συνάδελφο Λουί Γκρέχο ο οποίος ήθελε να παραστεί αλλά είναι αρρωστός και θα είχε πολλά σχόλια διότι είναι ένα θέμα που τον έχει απασχολήσει ιδιαίτερος. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι θεωρώ ότι η ιδέα αυτή είναι εξαιρετική, αλλά εγώ θα προτιμούσα εάν υπάρχει προακτική εξάσκηση νέων να γίνεται στη, στα θεσμικά όργανα και όχι στι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις σας ψάξουν τους δικούς τους υποψηφίους ε, για να κάνουν στάζ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε εμείς να φροντίσουμε για τους δικούς μας και αυτή είναι μία παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω. Έχω και μία δεύτερη ερώτηση σχετικά με τις 15 Οκτωβρίου που προβλέπετε. Ε, ε, αντιλαμβάνουμε ότι προβλέπετε μία πολύ μεγάλη εκδήλωση και χαίρεστε ότι θα σας διαθέσουμε την Ολομέλεια. Νόμιζα ότι θα κάναμε από κοινού κάποια εκδήλωση εξού και η διατύπωση κάποιος με ενόχλησε ή θα γίνει μία κοινή συνεδρίαση την οποία θα οργανώσουμε στην Ολομέλη αλλά τι προβλέπετε συγκεκριμένα δεν έχω ακούσει κάτι συγκεκριμένο επ' αυτού και με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι ένα θέμα όπου θα μπορούσαμε ε, να εμπλέξουμε και τους νέους αλλά καταλαβαίνω ότι η απονομή βραβείων είναι κάτι διαφορετικά, διαφορετικό. Πώς θα τα συνδέσουμε αυτά. Είναι μια ερώτηση που κατ' εμέ είναι πολύ σημαντική. Δεύτερον, γιατί δεν κάνουμε ένα κοινοβούλιο των νέων σχετικά με το θέμα αυτό. Για τους 20χρονους κάτι πιο μεγάλο, όπου οι ανταλλαγές μεταξύ νέων θα μπορέσουν να διεξαστούν σε ένα κοινοβούλιο όπου με το web stream που έχουμε θα μπορούν να συμμετάσχουν και μέσω του διαδικτύου νέοι από αλλού και να παρέμβουν περισσότεροι ε, επί του θέματος που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχω δει ε, να συζητείτε μέχρι στιγμή. Σήμερα το πρωί διαβάζοντας την εφημερίδα μου <clears throat> είδα κάτι πολύ ενδιαφέρον ότι εχθές στο κοινοβούλιο της Βάδης ε, Βουτεμβέργης ε, εορτάστηκαν ε, τα 60 χρόνια και εκτός από τις σημαντικές προσωπικότητες ήταν και δι, τρεις νέοι που είχαν προσκληθεί για να πούν τι είναι η Βάδη Βιντεβέργη και πώς εμπλέκεται η Ευρώπη στην περιφέρεια αυτή. Εν ώψη του τι πρόκειται να γίνει στις 15 Οκτωβρίου σας το αναφέρω και διαβάζω μία φράση από το άρθρο που μου άρεσε. Ένας από τους νέους που είναι φοιτητή νομικής είπε ότι η προοπτική των νέων είναι η Ευρώπη. Δεν είναι τόσο σημαντικά τα τοπικά σύνορα ακόμη και αν η τοπική προέλευση δεν εξαφανίζεται. Αυτό το λέει σαν ένας νοτιογερμανός. Ε, εάν λοιπόν υπάρχει κάτι τέτοιο νομίζω ότι είναι κάτι καλό και ε, έχω διάφορες ιδέες για το πώς μπορεί κανείς να βελτιώσει την εκδήλωση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι λόγω της οικονομικής ε, κρίσης είναι η σωστή στιγμή να εστιαστούμε ε, στην ανάπτυξη τη εσωτερική αγορά, διότι χρειαζόμαστε και οικονομική ανάπτυξη και νέε θέσει απασχόληση. Είναι λοιπόν η σωστή στιγμή για να κάνουμε διαφήμιση για την εσωτερική αγορά. Μ' αρέσει αυτή η ιδέα της ε, γενιάς του, του 1992. Κανένα πρόβλημα ποιοι θα είναι, πόσοι θα είναι οι αποδέκτες. Ε, πόσοι πόσους 20χρονους έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσους ε, θα ενδιαφέρει το θέμα. Αν έχουμε άμεση επαφή με τα πανεπιστήμια και τα σχολεία, ίσως είναι πιο εύκολο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τηλεόραση στις διαφημίσεις. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι την ε, ευρύτερη δυνατή υποστήριξη. Καλά και τα κοινωνικά ΜΜΕ, δεν τα χρησιμοποιώ εγώ βεβαίως, αλλά και δεν είμαι και ο μόνος. Αναρωτιέμαι πόσους 20χρονους μπορούμε να αγγίξουμε με αυτό το διαφημιστικό μήνυμα, την εκστρατεία, τη διαφημιστική για την εσωτερική αγορά. Years Αναρωτιέμαι αν ξέρουν ότι υπάρχει η εσωτερική αγορά όλοι αυτοί οι 20, 20χρονοι. Οι περισσότεροι, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρουν ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν επίτροπο και έναν βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολύ καλό θα ήταν ε, να εμπλακούν ε, οι νέοι, να τους πούμε, παραδείγματος χάρη, στη συνέντευξη ε, να τους κάνουν ερωτήσεις. Είχατε γεννηθεί όταν ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνειδητοποιήσουν ε, την ιστορία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Επίσης, άλλη ιδέα μπορούμε να εξετάσουμε είναι ένα είδος ε, μανιφέστου. Πώς θέλετε να είναι ο κόσμος το 2070, θα μπορούσε να τυκλοφορείτε το μανιφέστο να ε, χρησιμοποιήσουμε τη δημιουργικότητα των νέων, να φανταστούν σενάρια. Μπορεί και να μην ε, ε, υπάρχει ακόμη η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ αυτό προβλέπω πάντως. events foreseen in the Άλλα τώρα που προβλέπονται στα κράτη-μέλη, εκδηλώσεις στο διαδίκτυο, αυτό θα μπορούσε να αγγίξει πολλούς νέους. Επόμενη ομάδα η πράσινη δεν είναι ε, πλέον εδώ. Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που θέλει να σχολιάσει. Η κυρία Χάνσλικ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Κατ' εμέ, αυτό που λείπει είναι ισχυρή συμμετοχή από τη δική μας πλευρά, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί εμείς έχουμε επαφές και με τον ε, επιχειρηματικό κόσμο και με τον ακαδημαϊκό κόσμο. Θεωρώ ότι το κενό που εντοπίζω κατά κύριο λόγο είναι από δική μας πλευρά. Εμείς πρέπει να συμμετάσχουμε πιο ένεργα στην προώθηση α, της σημασίας της ενίας αγοράς είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσία της Ευρωπαϊκής και θα θέλαμε, αν είναι δυνατόν, να την ε, λάβουμε. Ε, δεν, εγώ δεν το πήρα το, το, το PowerPoint αυτής της παρουσίασης. Ίσως θα ήταν δυνατόν, Πρόεδρε, να μας διανεμηθεί. Γιατί και εμείς καλό είναι να προβληματιστούμε. Πώς μπορούμε να ε, καταστήσουμε κοινωνούς της όλης αυτής διαδικασίας τους 20χρονους ενιαία αγορά μπορεί να είναι και άγνωστη λέξη για τα πιο πολλά νέα παιδιά 20 ετών. Ε, άκουσα με προσοχή και προβληματισμό το λεγόμενο του κ. Μάντερς. Αυτά μπορώ να συμβάλλω και εγώ σήμερα μια συζήτηση. Θέλω να αναφερθώ σε ένα σέμα για να μπορέσετε να απαντήσετε σε όλα μαζί. Ε, μία συνάδελφος είχε πει ότι η διαφήμιση στα κράτη-μέλη θα ήταν καλή. Η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται ε, σε διαφημίσεις ε, για τα λουλούδια, για την πώληση του γάλακτος, για κάθε δυνατό κάτω από τον ήλιο. Οπότε θα μπορούσαμε και στο θέμα αυτό κάτι να προβλέψουμε και να αναφερθεί αυτό στην ομάδα εργασίας όταν θα υπάρχει μία μια συζήτηση. Ο κύριος Μάντερς ακόμη. Δεν είναι σοφότερο να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη που ζητούν ενισχύσεις να τους ε, υποχρεώσουμε, να τους, όχι να τους ζητήσουμε, να τους υποχρεώσουμε ένα μικρό ποσοστό των ε, διαφημίσεων ε, στην τηλεόραση να είναι μια μπλε οθόνη με τα αστεράκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν τους υποχρεώσουμε, εγώ ήμουν καλλιτέχνης στο παρελθόν και ξέρω ότι για όλα τα δημόσια κτιρία το 1% πρέπει να είναι για έκθεση αγαλμάτων και ε, πινάκων ζωγραφικής. Αυτό ήταν πολύ καλό για τους καλλιτέχνε. Γιατί να μην κάνουμε κάτι αντίστοιχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Yeah. Ευχαριστώ. Το έχουμε και στη Γερμανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο και πριν ε, ε, απαντήσετε έχει η Ρόζα το λόγο. Ε, θέλω να τοποθετηθώ και πάλι για αυτά τα στάζ ε, της περίπτωσης Πώς γίνεται να προτείνετε εσείς περίπτωση μαθητείας από κομισιών στο Κοινοβούλιο. Μήπως να ζητήσετε από εμά ε, που όσοι ενδιαφερόμαστε να δημοσιεύσουμε έναν κατάλογο, να προβούμε σε μια δήλωση για πρόσκληση ενδιαφέροντος. Ε, στο κάτω-κάτω αν είναι κοινή η εκδήλωση, είναι κοινό το event, να συμμετάσχουμε πιο ενεργά. Λοιπόν, κύριε Ντέριγκ, είναι common event, κοινό, κοινή εκδήλωση. Ε, Βεβαίω. Ευχαριστώ για όλε τι ερωτήσει, γιατί μπορώ να διευκρινίσω κάποια πράγματα, αλλά και να πάρω και κάποια ω τροφή για σκέψη και για μένα. Σε ό,τι αφορά την προώθηση, τώρα ξεκινούμε την εκστρατεία στα κοινωνικά μέσα στο διαδίκτυο. Άρα λοιπόν χρειάζεται πολλή δουλειά και εσεί μπορείτε να συμμετάσχετε ενεργά και επικοδομητικά. Κατά πόσον θα υπάρχουν ε, τηλεοπτικά σποτ θα το δούμε, γιατί είναι πολύ δαπανήρη μια τέτοια εκστρατεία. Θα το δούμε. Ακούσα ε, όμως πολύ χρήσιμες ε, προτάσεις. Ίσως κάτι από αυτό να γίνει πραγματικότητα. Πάντως, εργαζόμαστε εντατικά με τους εταίρους μας. Ήδη έχουμε περίπου 200 οργανώσεις εταίρους που είναι από αγροτικές ενώσεις νεολαίας μέχρι πανεπιστημιακές, ε, φοιτητικές ε, οργανώσεις, από κλαδικές ενώσεις, από το φαρμακευτικό κλάδο, την, τις ε, κοινωνικές επιστήμες κτλ. κτλ. οργανώσεις που εκπροσωπούν τους νέους ανέργους, οργανώσεις που στηρίζουν νέους επιχειρηματίες. και αυτό που κάνουμε αυτήν την εκστρατεία είναι ακριβώς να εντοπίσουμε τους νέους ενήλικες που συμμετέχουν σε αυτές τις οργανώσεις για να ακούσουμε τη δική τους οπτική γωνία. Τώρα για τις ε, κεντρικές εκδηλώσεις, τα κεντρικά event, θα τα ξανασυζητήσουμε σε αυτή την Διευθύνουσα Επιτροπή, ένα steering committee που έχουμε δημιουργήσει από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε ευχαριστούμε και πάλι για τη συμμετοχή. Πράγματι, αυτές οι εκδηλώσεις είναι κοινέ, είναι κοινό event. Και βεβαίω η βράβευση θα γίνει κατά τη διάρκεια τη κύρια εκδήλωση και αυτό θέλουμε να είναι μια πολύ δυναμική εκδήλωση και ανατριπτική, αν θέλετε, να ξεφεύγει από τα τετριμένα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, και έχετε δει και πρέπει να βρούμε κάποια links, να, δούμε πώς θα διασυνδέσουμε αυτή την εκστρατεία με, με πολλά μέσα, τα μέσα ενημέρωσης και με πολλούς τρόπους το κατά πόσον δεν έχουν ιδέα πολλοί νέοι για την ενιαία αγορά. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κάποια εκατομμύρια νέοι είναι εκεί έξω που δεν έχουν ιδέα για την ενιαία αγορά. Σε ένα βαθμό αυτό το project με τους λίγους πόρους που έχει προσπαθεί να αντιμετωπίσει και αυτό το πρόβλημα με το ίντερνετ και τη διάδραση. Ελπίζουμε να ε, διδάξουμε κάποια πράγματα, αλλά όχι να διδάξουμε από, ε, την έδρα, αλλά να τους προσελκύσουμε αν θέλετε. Η μαθητεία, τα στάζ θα αφορά και επιχειρήσεις με κάποια φήμη, επιχειρήσεις ε, ε, των ε, ΜΜΕ. Αλλά θεωρούμε ότι αν συμμετάσχει στα, στην προοπτική της μαθητείας και του Προκοινοβούλιο θα είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Προσβλέπω σε επικοδομητική συζήτηση και τους επόμενους μήνες. Όπως είδατε υπάρχουν πολλές προτάσεις και υποθέτω ότι το θέμα αυτό εν πάση περιπτώσει θα συζητηθεί πριν από το καλοκαίρι θα το ξανασυζητήσουμε για να μας πείτε πού βρίσκεστε ε, και κατά τρόπον ώστε μέχρι τις 15 Οκτωβρίου να μπορέσουμε να συμβάλλουμε με προτάσεις. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μάντερς. Ευχαριστώ συνήθως ορίζουμε ημερομηνία, καταλεκτική ημερομηνία για τροπολογίες. Μπορούμε να το κάνουμε και γι' αυτό. Υπάρχει μια ομάδα εργασία Τόνι, και υποθέτω ότι εκεί θα συμμετέχει και ένας φιλελεύθερος. Και αυτή συναλλάσσεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, είδα ότι εσεί είσαι στην ομάδα εργασία και κατά δεύτερον λόγο το θέμα αυτό ε, θα τεθεί στην ημερήσια μας διάταξη για να παρουσιαστεί ε, και αυτό θα γίνει αύριο, θα γίνει ένα πρωινό στις 10 για να παρίστανται όλοι. Και τώρα απλώς πρέπει να σας πω πότε είναι η επόμενη συνεδρίαση, 3η 8 Μαΐου όλη την ημέρα και σας εύχομαι μια υπόλοιπη καλή πέμπτη.